Λοιπόν, καλημέρα σας. Σας προτείνω να αρχίσουμε τις εργασίες μας. Ε, ε, λοιπόν, ε, πραξικόπημα επειδή αποουσιάζει έτσι για πάρα πολύ λίγο και δικαιολογημένα η πρόεδρός μας, καλούμε να προεδρέψω εγώ. Ε, και την αντιπρόεδρη επίσης. Και σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες του Κοινοβουλίου, τον ιστορικό μας κανονισμό, ε, προεδρεύει ο πρεσβύτερος, παρακαλώ, που φυσικά είναι ο συνάδελφος Έλμαρ Μπρόκ. ο οποίος από τις συνθήκες έχει παρακολουθήσει από τη συνθήκη της Ρώμης ε, ε, αλλά ε, κολλείεται σήμερα το πρωί και αμέσως μετά τον Έλμαρ είμαι εγώ ο πρεσβύτερος. Πρέπει να σας πω ότι με ανάκτημα ε, ανάμεικτα συναισθήματα προεδρεύω. Ε, θα ήθελα να μπορώ να προεδρεύω για άλλους λόγους από την ηλικία μου. Εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ και να ε, διαχειριστώ την προεδρία. Αν δεν διαφωνείτε προχωρούμε έτσι. Πρώτο σημείο στην μέση διάταξη, έγκριση αυτή. Δεν ξέρω αν έχετε σχόλια και παρατηρήσει, αλλιώ θεωρείται εγκεκριμένη. Στη συνέχεια, ανακοινώσεις του Προέδρου. Έχουμε βασική ανακοίνωση, πέρα από το γεγονός ότι ε, ε, μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μα, Δεν βλέπετε τι κάμερε, αλλά από ό,τι φαίνεται ο κόσμο ολόκληρο, έχει στραμμένα τα μπλέμματά του και τα αυτιά του εδώ. Η βασική ανακοίνωση είναι η κατάσταση του τριμερίου διαλόγου σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Είναι εδώ ο εισηγητή μα, ο Γιώργη Σόπφλιν και θα προτείνω να μα κάνετε μια σύντομη παρουσίαση ε, για αυτή την υπόθεση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πώς έχει η κατάσταση των πραγμάτων τώρα κάπως δύσκολη θα τη χαρακτήραζα αυτή τη στιγμή. Ακόμα δεν έχουμε κοινή θέση με τους υπόλοιπους και εισηγητές. Η εμπλοκή έχει να κάνει με την ηλικία των υπογραφών. Μπορεί να υπογράφει κάποιος από την ηλικία των 16 ετών. Ε, εμείς ε, λέμε ναι, ε, τα κράτη-μέλη μπλοκάρουν, η Προεδρία ε, το κοιτάει. Ε, την άλλη εβδομάδα υπάρχει τριμερής διάλογος και είναι την ίδια ώρα με τις ψηφοφορίες την Τετάρτη το απόγευμα στις 5. Θα δούμε πώς θα το ρυθμίσουμε. Δεν μπορώ να σας πω πολλά περισσότερα. Δεν είμαι 100% αισιόδοξο αν μπορώ να το πω έτσι. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο αν δεν αλλάξουν την εντολή μου, δηλαδή η πλειοψηφία ε, ζητεί να είναι η στάνταρ ηλικία 16 ετών, τα κράτη-μέλη ούτε να τα ακούσουν. Αν δεν αλλάξει η κατάσταση θα πάει στη Ρουμανική Προεδρία το θέμα. Ελπίζω την άλλη φορά να σας έχω καλύτερα νέα. Καλώς, ευχαριστώ αγαπητές συνάδελφοι. Καλά, κανονικά, ε, καταρχήν η Αυστριακή θα πρέπει να είναι υπέρ, γιατί νομίζω ότι είναι η μόνη χώρα όπου ψηφίζει κανείς από την ηλικία των 16 ετών. Και η Μάλτα. Α, και η Μάλτα, μάλιστα. Ωραία. Ο Γιώ Λάινεν. Στα αγγλικά. Α, στα γαλλικά, με πώς θες να τα πω γαλλικά. Ε, ε, στα γαλλικά. Αυτή ήταν η απόφαση μας, να μπορούν να συμμετέχουν και οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που δεν είναι νομοθετικού περιεχομένου, εκφράζει ο κόσμος την άποψή του. Και, ε, και δική μας επιθυμία είναι αυτή ακριβώς να συμμετέχουν οι νέοι. Θα πρέπει να βρούμε κάποια λύση. Υποχρεωτικό δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε, γιατί μόνο η Μάλτα και η Αυστρία έχουν δικαίωμα ψήφου ε, στην ηλικία των 16 ετών, πολιτική ενηλικίωση δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, αλλά μπορούμε να εκφράσουμε εμείς την επιθυμία μας, όλο και περισσότερο ή όλο και περισσότερα μέρη να δεχθούν την ηλικία των 16 ετών. Εγώ δεν έχω χάσει κάθε ελπίδα, διατηρώ τις ελπίδες μου να ολοκληρωθεί αυτό το θέμα στην Αυστριακή Προεδρία. Ο κύριος Σόφιν, μακάρι να συμμεριζόμουν το δική σου αισιοδοξία, γιατί Ακούω ότι φρονούν τα κράτη-μέλη, όχι η Αυστριακή Προεδρία, το βλέπει πολύ θετικά και το υποστηρίζει. Με το που θα δουν κάποια κράτη-μέλη το 16 είναι κόκκινη γραμμή, να μην πω κόκκινο πανί. Και υπάρχει ε, πλειοψηφία που μπορεί να μπλοκάρει, ανασταλτική πλειοψηφία, στο, ε, μια ψηφία συγγνώμη, στο Συμβούλιο. Ε, δεν θέλουν ούτε να τα ακούσουν αυτό το θέμα της ηλικίας των 16 ετών. Πολύ ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Και σημειώνω ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα χρονικό ημερομηνίας και ώρας για τον προσεχή τριμερή διάλογο. Διότι γνωρίζετε αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή τελειώνει η θητεία τώρα, χρειαζόμαστε ε, χρονοθυρίδες για ψηφοφορίες επιπλέον των μεσημβρινών. Και την άλλη εβδομάδα, την Τετάρτη το απόγευμα, έχουμε έκτακτη ώρα ψηφοφορίας στις 5 το απόγευμα και παρακαλώ να ε, προετοιμαστείτε. Ωραία. Προχωρούμε στο σημείο 3. Μετά τη συνέδριαση των συντονιστών, και με γραπτή ε, διαδικασία αποφάσισαν να συσταθεί ομάδα εργασίας της ΑΦΚΟ για το Brexit, ε, όπου θα συμμετέχουν η Πρόεδρος, ο εισηγητής και οι Σκιώδης. Οι συντονιστές συμφώνησαν ε, να οριστεί η εισηγητής ο Γκίφερ Χόφστατ και οι Σκιώδης θα είναι από το ΕΛΚΟ Ελμαρ Μπρόκ, προφανώς, από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη, από τους συντηρητικούς ο Μόρτεν Μέσερ Σμίτ, αντιπρόεδρος μας, από την Γκου η Γκάπη Τσίμερ, από τους πρασίνους ο ίδιος ο Φίλιπ Λαμπέρτς, από το EFTD ο Μπάτεν και ε, από το ENF ο Χέρολφ Άνεμανς. Έτσι, αυτό αποφάσισαν οι συντονιστές. Αν δεν διαφωνείτε, την εγκρίνουμε. Alors, Και ερχόμαστε στο σημείο 4, που είναι η έκθεση του Πάολο Ρανζέλ για την τροποποίηση της απόφασης του Κοινοβουλίου σχετικά με το καθεστώς του διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του. Πάολο, μπορείς να μας δώσεις τα φώτα σου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά από μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Οράιλη, πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, η Επιτροπή μας ε, ξεκίνησε μια συζήτηση για την παρουσίαση της μελέτης των κανονισμών και των γενικών προϋποθέσεων που διέπουν τα καθήκοντα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβήτη και της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας και των σχετικών καθηκόντων τους. Έχει έρθει η ώρα να παρουσιάσουμε το σχέδιο έκθεσης, το οποίο είναι κάπως ιδιαίτερο από θεσμική άποψη. Όπως γνωρίζετε, αποτελεί δικαίωμα πρωτοβουλίας ε, του Κοινοβουλίου, κάτι σπάνιο. Επίσης, ε, είναι ιδιαίτερη έκθεση και διαδικαστικά. Όχι μόνο περιλαμβάνει μια σειρά πολιτικών κατευθύντηρων γραμμών, αλλά και το νέο καθεστώς της διαμεσολαβήτριας και διαμεσολαβήτη. Θα λέγαμε αμερόληπτος, ουσιαστικά μη δικαστικός πάροχος δικαιοσύνης. Έχει πέρασει μία δεκαετία μετά από την τελευταία τροπολογία του σημερινού καθεστώτος. Στο μεταξύ, τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να επικαιροποιηθούν οι διατάξεις ώστε να επιτευχθεί πλήρη συμμόρφωση με το νέο θεσμικό πλαίσιο και συνταγματικό πλαίσιο της Ένωσης. Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε πώς θα πάμε σε εκλογές χωρίς να έχουμε ένα καθεστώ για τον δημοσιολαβητή το οποίο να σύμφωνει με τις συνθήκε τη Λισαβόνα. Το σημερινό καθεστώ λοιπόν θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με ένα νέο κανονισμό σύμφωνα με τι συνθήκε. Πέραν από την επικαιροποίηση των διατάξεων του καταστατικού, το σχέδιο ε, προωθεί και μία ε, εξέλιξη συνέχεια που καλύπτει δύο δεκαετίες δραστηριοτήτων του Δημοσιολαβητή με όλο ένα και πιο αυξημένη προβολή μεταξύ του κοινού, των οργανισμών, των θεσμών ε, συχνά ακολουθούν τις συστάσεις ε, του Δημοσιολαβητή εθελοντικά. Αποτελεί μια ηθική μορφή για τους Ευρωπαίους πολίτες ε, είναι ο επόπτης ως Ευρωπαϊκή Αρχή είναι μέσα στο σύστημα και ταυτόχρονα από πάνω του χρησιμοποιεί ήπια αλλά ε, δύναμη αλλά, και εξουσία αλλά μεγάλης επιρροής. Οπότε θέλω να τονίσουμε πόσο σημαντικός είναι ο δημοσιολαβητής και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του ως ήπια εξουσία στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. οι αρμοδιότητες του ή της ε, είναι ήπιες, ήπιας μορφής. Ο ρόλος αυτός απαιτεί συνταγματική και νομοθετική αναγνώριση της αυτονομίας ταυτόχρονα με τα απαραίτητα εργαλεία για την εκτέλεση των καθηκόντων. Λοιπόν, αμεροληψία, ανεξαρτησία, ουδετερότητα, αυτονομία. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά φυσικά του Δημοσιολαβητή. Ταυτόχρονα πρέπει να παρέχουμε στον Ευρωπαίο Δημοσιολαβητή τα μέσα, τα εργαλεία, ώστε να μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Αυτή την ισορροπία προσπαθούμε να την ε, επιβεβαιώσουμε τονίζοντας ότι όχι μόνο κάθε οργανισμός και κάθε θεσμικό όργανο πρέπει να έρχεται σε επαφή με το δημοσιολαβητή αλλά και ότι ε, πρέπει ο διαμεσολαβητής να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες, έγγραφα, μαρτυρίες, ώστε να μπορεί να χειριστεί καταγγελίες και να πραγματοποιεί έρευνες και ε, παρακολούθηση των ερευνών με δική του πρωτοβουλία. Πρέπει λοιπόν να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες. Ε, όσον αφορά τώρα μια συστημική προσέγγιση προς το κείμενο, θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντική είναι η σχέση μεταξύ δημεσολαβητή και άλλων ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών. Στο σχέδιο έκθεσης, η πρώτη ετήσια έκθεση ε, απαιτεί παρουσία στο κοινοβούλιο, κοινοποιεί το, την Ευρωπαϊκή Συγγελία για ποινικά δικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και συνεργάζεται με, οργανισμούς, με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με ίδιο τύπο αρχές στα κράτη-μέλη. Υπάρχει αυτό το τρίγωνο λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τέλος, ως τελευταίος πυλώνας του σχεδίου έκθεσης, το ελάχιστο περιεχόμενο των εκτελεστικών διατάξεων που θα υιοθετούνται από το δημοσιολογητή τώρα πρέπει να διευκρινιστούν. Αυτό το ελάχιστο περιεχόμενο περιλαμβάνει σε αυτή την εκδοχή του κειμένου τα διαδικαστικά δικαιώματα του καταγγέλλοντος και του θεσμού, οργανισμού, γραφείου, τη διεκπαιρέωση και το κλείσιμο μιας καταγγελίας και την ίδια πρωτοβουλία και τις ε, έρευνες ε, συνέχειας και τις ε, σχετικές προφορίες. Έτσι πιστεύω ότι η επιτυχία αυτής της νομοθετικής διαδικασίας θα εξαρτήσει σε μεγάλο βαθμό από το πώς εμείς ως μέλη της Επιτροπής μπορούμε να συμπεριλάβουμε χωρίς να ζημιώσουμε. Αυτό ουσιαστικά είναι ο βασικότερος στόχος, να βελτιώσουμε χωρίς να καταστρέψουμε. Έχουν περάσει σχεδόν δύο θητειε μετά από τη Λισαβόνα και σίγουρα οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θέλουν να παραμείνει απερχαιωμένο το καταστατικό για μια τέτοια μορφή όπως η τη. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν να έχουμε ένα νέο κανονισμό και τις γενικές ε, προποθέσει που διέπουν το καθεστώς του διαμεσολαβητή. Ωστόσο θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφή σε ένα πράγμα, όχι με εκβάθρον μεταρρύθμιση. Αντιθέτω με ε, επικύρωση και ανάδειξη του ε, συνταγματικού ρόλου αυτής της μορφής. Εξουσία του είναι να μην έχει εξουσία. Έχει συνταγματικό ρόλο να διασφαλίζει ότι όλοι συμμορφώνονται με αυτόν. Αυτοί είναι οι πέντε πυλώνες του σχεδίου και είμαι έτοιμος να ακούσω τις επικρίσεις και τα σχόλιά σας. Euh, Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Σαφέστατη παρουσίασή σα αυτή. Πρόκειται για μια διαδικασία τελείω ασυνήθιστη που θα θέλαμε να δούμε να εφαρμόζεται κι αλλού όπου η νομοθετική πρωτοβουλία εναπόκειται στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή, επί της ουσίας, αρμόδια είναι η δική μας Επιτροπή. Και ε, επιλαμβάνεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωμοδοτεί και το Συμβούλιο στη συνέχεια ψηφίζει. Ούτε καν ψηφίζει, συνενεί. Demande si du côté... Euh, λοιπόν, οι πολιτικές ομάδες θέλουν το λόγο. Σοσιαλιστές, Ενρίκη Γκερέρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Ρανζέλ. Βλέπω βλέπετε πόσο ενδιαφέρονται οι δικοί μου συνάδελφοι περισσότερο από τους δικούς σας και υπάρχει και η βυρική αλληλεγγύη που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα αυτό και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ρανζέλ που σκέφτεται να ε, εντάξει ε, ορισμένα στοιχεία που προτείναμε εμείς, η δική μας πολιτική ομάδα. Συμφωνώ απολύτως με τις τρεις βασικές γραμμές της επιχειρηματολογίας σας. Πρώτον, επειδή έχουν περάσει 20 χρόνια και έχει εγκριθεί και η συνθήκη της Λισαβόνας και μερικές άλλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις έχουν μεσολαβήσει, ε, πρέπει να προσαρμοστεί και το καθεστώς που διέπει τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις κανονιστικές και μέχρι και συνταγματικές αλλαγές που έχουν μεσολαβήσει στην περίοδο αυτή. Αυτή θα ήταν ε, η πρώτη γραμμή. Η δεύτερη γραμμή που αναπτύξατε είναι εξέλιξη, ε, συνεχεία όμως, δηλαδή βελτιώνουμε όπου μπορούμε ε, τους όρους και τρόπο εργασίας ε, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα θα πρέπει να έχουν ένα σεβασμό και να μην ε, επεμβαίνουν και παρεμβαίνουν παρά μόνο για λόγους πληροφοριακούς. Όλα αυτά για να υποστηρίζουν το έργο του διαμεσολαβητή και χωρίς να αλλάξει ε, φύση ε, το θεσμικό όργανο και να μην υπάρξει καμία ανισορροπία στις σχέσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Εν όψη πιο βαθιών αλλαγών, ας πούμε, μέσω πρόθεσμα. Όταν θα γίνουν πιο βαθιές αλλαγές, αυτό θα το ξαναδούμε. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ουσιαστικές. Και το τρίτο που είπατε, και ε, μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό είναι το εξής. Ε, μ' αρέσει καλύτερα όρος που χρησιμοποιείται στα πορτογαλικά. Ε, κάποιος που ε, παρέχει δικαιοσύνη αλλά σε εξοδικαστική οδό. Μ' αρέσει αυτό. Να μην πούμε σε κάτι που προτάθηκε από άλλους, ε, δηλαδή να έχει τη δυνατότητα ο διαμεσολαβητής να ε, μπορεί να ε, επεμβαίνει και ε, να είναι τμήμα της διαδικασίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν μ' αρέσει αυτό. Η εξουσία του είναι ε, ακριβώς ότι δεν έχει εξουσία, όπως είπατε στο τέλος, αλλά ε, έχει ένα ηθικό κύρος και ανάστημα, οπότε δεν μπορεί να είναι ένας διάδικος, ας πούμε, σε μια ε, μακροματική διαδικασία στο δικαστήριο. Βεβαίω, οι εξουσίε και οι αρμοδιότητε μπορούν να βελτιώνονται με την υλικοτεχνική υποδομή, βελτίωση των πόρων, οικονομικών, ανθρώπινων κλπ. Αλλά και με κάποιες καινοτομίες ε, που έχουν προκύψει ας πούμε από τη δημιουργία του, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και πάλι αυτό που χρειάζεται ο διαμεσολαβητής είναι περισσότερη πληροφόρηση από τα θεσμικά όργανα. Επίσης είναι καλό να ενισχυθούν οι σχέσεις με τους εθνικούς διαμεσολαβητές και συνήγορους του πολίτη σε χώρες μέλη. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε να έχουν ε, αντικρουόμενη δράση, κυρίως ε, λόγω έλλειψης συνεννόησης, ε, επικοινωνίας και πληροφόρησης. Και τέλος στην πρότασή σας υπάρχει κάτι που μου φαίνεται σκόπιμο. Ο διαμεσολαβητής μπορεί ο ίδιος να ζητήσει να έρθει σε, ενώπιον των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που χειρίζονται θέματα σχετικά με παράπονα και καταγγελίες που έχει λάβει ο διαμεσολαβητής από τους πολίτες. Είτε να είναι παρόν στη συζήτηση, είτε να τους διαβεβάζει κάποια αιτήματα. Δηλαδή να μην το ζητάμε εμείς να έρθει, ε, να έχει τη δυνατότητα ο διαμεσολαβητής ή η διαμεσολαβήτρια να ζητήσει από την εκάστοτε επιτροπή να δεχτεί την παρουσία του. Την παρουσία της. Οπότε κύριε Ρανζέλ, εμείς δεν θα σας κάνουμε κανένα κατάλογο τροπολογιών. Μπορεί. Πολύ λίγες, αν χρειαστεί, θα το σκεφτούμε. Μια-δυο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητοί συναδελφοί. Λοιπόν για το ECR ο Ισκιώδης Μόρτερ Μέσερ Σμιτ δεν είναι εδώ. Υπάρχει κάποιος άλλος για να μιλήσει εκ μέρους του ECR. Δεν βλέπω. Για το Aldo Μάιτε Πάγκα Ζαορτουντόα, δεν τη βλέπω. Για τους πράσινους Ιωσέπ Μαρία Τρικάβρας. Βλέπω ότι οι Ισπανοί συνάδελφοι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτό το σημαντικό θέμα, αλλά δεν είναι παρόντες. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο, Κατσδιάη. Ζόρζι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η έκθεση, ιδιαίτερα για τους ε, μη δικαστικούς παρόχους ε, δικαστικό, υπηρεσιών δικαιοσύνης. Με ενδιαφέρει πολύ ο θεσμός του διαμεσολαβητή, της διαμεσολαβήτριας. Θα έπρεπε να είναι ουδέτερη η περιγραφή, τέλος πάντων. Υπάρχει τέτοιος ε, θεσμός ε, σε όλα τα κράτη-μέλη ή υπάρχουν κάποια που δεν έχουν διαμεσολαβητή. Θα ήταν ενδιαφέρον για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Επίσης, υπάρχει σχέση μεταξύ του διαμεσολαβητή και των διοικητικών δικαστηρίων. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια του κυρίου Γκερέρο Σαλόμ και του κυρίου Σόπφλιν, επί του συντονιστή. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι προσπάθησα να κοιτάξω τον όρο διαμεσολαβητής ombudsman. Είναι σουηδική λέξη. Κοίταξα λοιπόν να δω αν είναι αρσενικού γένους ή θηλυκού, αλλά είναι ουδέτερο. Δεν είναι τόσο εύκολο να σας το εξηγήσω. Και εσείς το ξέρετε καλύτερα γιατί η γλώσσα σας είναι αρκετά δύσκολη. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και μετά από συζητήσεις με συναδέλφους, ο θεσμός εκλαμβάνεται, η θέση εκλαμβάνεται ως ε, θέση ενός προσώπου, όχι άντρα-γυναίκας. Τώρα το man ακούτε, σκέφτεστε αγγλικά και νομίζετε πως είναι άνδρας. Δεν είναι όμως έτσι. Έπειτα. Σχεδόν όλες οι χώρες, ε, από όσο γνωρίζω, έχουν αυτόν τον θεσμό. Και γίνονται κοινέ συναντήσεις, ανταλλάσσονται απόψεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όπως γνωρίζετε γίνεται αυτό και στα συνταγματικά δικαστήρια της Ευρώπης. Υπάρχει συνεργασία με τον διαμεσολαβητή. Υπάρχει λοιπόν μια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, μια σύγκριση σε εθνικό επίπεδο. Το δίκτυο αυτό είναι ανεπίσημο, οπότε δεν έχει επίσημη καθορισμένη δομή. Είναι μια συνάντηση έτσι ώστε να γίνεται αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών. Έπειτα δεν υπάρχει σχέση με κάποιο συγκεκριμένο τύπο δικαστηρίου. Όπως γνωρίζετε, πολλές καταγγελίες έχουν ε, διοικητικό περιεχόμενο. Θα μπορούσα ε, λοιπόν μια τέτοια καταγγελία να πάει σε ένα ε, διοικητικό δικαστήριο. Όμως, όπως γνωρίζετε, τα δικαστικά συστήματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Πολλές ε, χώρες έχουν ένα συγκεκριμένο ε, παράρτημα, άλλες έχουν ξεχωριστό δικαστήριο εντελώς. Και φυσικά δεν κινδυνεύει ο θεσμός του διαμεσολαβητή, όμως σε εθνικό επίπεδο ο διαμεσολαβητής έχει αρκετά καθήκοντα, βέβαια δεν μπορεί να ασχοληθεί με ποινικά ζητήματα. Και αν και αν είμαστε έτσι πολύ δογματική. Δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στο σοφρονιστικό σύστημα και τον θεσμό του διαμεσολαβητή. Αυτά είναι αρμοδιότητα των ποινικών δικαστηρίων σε περίπτωση που έχει προκύψει κάποια καταγγελία ποινικού χαρακτήρα. Όμως όπως τόνισε και ο Ενρίκε Γκερέρο, είναι σημαντικό ο διαμεσολαβητής να μην εμπλέκεται σε δικαστικά ζητήματα. Διότι είναι διαμεσολαβητής ακριβώς και δεν έχει δικαστικές αρμοδιότητες. Δεν δικάζει εγκληματίες, δεν συμμετέχει καθόλου σε αυτήν την διαδικασία. Τώρα βέβαια, υπάρχει η δυνατότητα ο διαμεσολαβητής να διεξάγει μια έρευνα που έχει μεν ε, σχέση με μια δικαστική υπόθεση χωρίς να είναι αμυγός ε, τέτοια, δηλαδή μια έρευνα για ένα διοικητικό θέμα ή για ε, εργασιακές σχέσεις. Όπως γνωρίζετε, για τα εργασιακά ζητήματα δεν είναι η τελευταία λύση ο διαμεσολαβητής, διότι διαφορετικά θα κατακλυζόταν από τέτοιου τύπου καταγγελίες. Έχουμε ζητήσει λοιπόν να εισαχθεί μια ρήτρα όπου η προσφυγή στο διαμεσολαβητή θα είναι μόνο ε, η έσχατη λύση. Και φυσικά δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν και δικαστήρια για τέτοιου είδους υποθέσεις. Τέλος, να σας πω ότι στα πορτογαλικά η μετάφραση του διαμεσολαβητή Ombudsman μεταφράζεται ως πάροχος δικαιοσύνης κατά λέξη, διότι δεν χρησιμοποιείται ε, μόνο σε δικαστικό πλαίσιο, είναι πάροχος δικαιοσύνης, δημιουργεί δικαιοσύνη. Αυτό είναι ε, το όνομα του διαμεσολαβητή στα πορτογαλικά και έχουμε επιλέξει αυτή τη διατύπωση ακριβώς για αυτές τις ε, μικρές λεπτομέρειες που δίνουν αυτήν την ε, μη δικαστική διάσταση στις δραστηριότητες του διαμεσολαβητή. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Στην περίπτωση της Γαλλίας, Εκεί έχουμε αυτό που ονομάζουμε διαμεσολαβητή της δημοκρατίας, αλλά και έναν υπερασπιστή δικαιωμάτων, που είναι ένας από τους παλιούς μας συνάδελφους ο Ζακτυμπό, αυτή τη στιγμή. Κάθε υπουργείο καλείται να δημιουργήσει τον δικό του διαμεσολαβητή. Το πρόβλημα που αναφέρεται πιο συχνά στη Γαλλία έχει να κάνει ε, στις σχέσεις με τις φορολογικές αρχές ε, οι οποίες είναι κακές και που οδηγούν τους Γάλλους ε, στο να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους απευθείας χωρίς κανένα διαμεσολαβητή. Αλλά ο θεσμός υφίσταται. Και εμπνέεται και από τι ιδιότητε του Ευρωπαίου Δημοσιολαβητή, ειδικότερα όταν βελτιώθηκε όπω θα βελτιωθεί από τα όσα προτείνει ο εισηγητή μα ο κ. Ραγκέλ και οι τροπολογίε των σκιωδών. Προβλέπετε ότι οι προθεσμοί για τι τροπολογίε είναι η 13η Δεκεμβρίου στι 5 το απόγευμα, την επόμενη εβδομάδα. Πρέπει να εγκρίνουμε την ε, εκθέση στις 22 Ιανουαρίου και η Ολομέλεια θα την εγκρίνει την εβδομάδα 11 με 14 Φεβρουαρίου. Σας προτείνω τώρα να περάσουμε στην έκθεση της Mercedes Μπρέσου. Αφορά την εφαρμογή των διατάξεων των συνθήκων σχετικά με την εξουσία του Κοινοβουλίου για άσκηση πολιτικού ελέγχου επί της Επιτροπής. Mercedes, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, τώρα θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. Ε, το συζητήσαμε ήδη την προηγούμενη φορά για τη δομή της έκθεσης. Έχουμε λάβει 86 τροπολογίες και μια γνωμοδότηση της, επιλογής, της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Θα ξεκινήσω από αυτήν. Υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις. Πιο συγκεκριμένα, σε τελική ανάλυση συμφωνούν με την έκθεση υπενθυμίζουν ότι το 80% της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης αποτελεί το αντικείμενο κοινή διαχείρισης με τα κράτη-μέλη. Εκεί τίθεται λοιπόν ένα πρόβλημα, απαιτείται πιο καλό συντονισμός μεταξύ Κοινοβουλίου και Εθνικών Αρχών Ελεγκτικών. Ο συντονισμός αυτός έχει κάποια κενά, διότι μερικές φορές ε, οι εθνικές αρχές ε, δεν είναι διατεθειμένες ε, να λάβουν υπόψη τις συστάσεις ή να πραγματοποιήσουν τις έρευνες ε, που ζητά το Κοινοβούλιο. Η γνωμοδότηση λοιπόν αυτή επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης ε, σε θέματα πολιτικού ελέγχου της Επιτροπής διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι το μόνο επιπεδης διακυβερνησης σε θεματα πολιτικου ελεγχου της επιτροπης διοτι όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. θέλει λοιπόν αυτό το πρόβλημα κυρίως κατακόρυφα, περισσότερο από τη οριζόντια. Οι τροπολογίες λοιπόν όπως είπα ήταν 86. Το σημαντικότερο θέμα στο οποίο επικεντρώνονται οι τροπολογίες είναι η επιλογή και ο έλεγχος ε, του Γενικού Γραμματέα της Κομισιόν και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αυτά, οι ανησυχίες που αφορούν τις εξουσίες ε, της Κομισιόν όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις και τις κατεξιδότητες πράξεις και οι δυνατότητες ελέγχου του Κοινοβουλίου, το ζήτημα της ε, σπουδαιότητας της διαδικασίας του κορυφαίου υποψηφίου του Spitzenkandidat το πώ θέλουν να ενισχυθεί και να διατηρηθεί αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν πολλέ τροπολογίε γι' αυτό. Επίση, είχαμε τροπολογίε κατά τη ιδέα ε, μείωση του κατοφλίου για του ορίου για την πρόταση μομφή. Αυτό θα απαιτήσει πολλή δουλειά με τους κοιόδης φυσικά. Επίσης, ε, περιλαμβάνεται η ιδέα χαλάρωσης ε, ε, της ιδέας ε, ανάθεσης ευθύνης στους επιτρόπους ζήτησε, απέτησε να λογοδοτούν οι επίτροποι. Επίσης υπάρχουν πολλές τροπολογίες για τις αυξημένες ευθύνες και λογοδοσία των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα το συζητήσω τώρα. Αυτό είναι σημαντικό κομμάτι και της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ελεκτού Προϋπολογισμού. Άλλες τροπολογίες υπάρχουν επίσης, ε, για παράδειγμα, σε σχέση με το είναι αναφορά εντό τη έκθεση για το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και εκεί, όπω ξέρετε, πάντα εκφράζεται κάποια ανησυχία όσον αφορά το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων περιφερειακών κοινοβουλίων. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά περιφερειακά κοινοβούλια, περιφερειακά συγγνώμη, όχι εθνικά, ε, υπάρχουν περιφερειακά κοινοβούλια που πρέπει να εφαρμόσουν τους κανόνες ε, υιοθέτησης ευρωπαϊκών, ε, ευρωπαϊκής θετική εξουσία. Και εκεί υπάρχει μια εκτελεστική εξουσία που μας διαφεύγει σχεδόν απόλυτα. Και αυτό το ζήτημα λοιπόν χρήζει εξέτασης. Ε, στις συμβαστικές τροπολογίες. Το επόμενο μας βήμα είναι η συνεδρία των σχεδόν εισηγητών την οποία ελπίζω να μπορούσα να οργανώσω στο Στρασβούργο όχι σε αυτό το Στρασβούργο, στο επόμενο του Ιανουαρίου. Τετάρτη 16 Ιανουαρίου ελπίζω και πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην επιδίωξη συμβιβασμών σε τέσσερα σημεία τα, που είναι τα πιο ευαίσθητα, τα πιο περίπλοκα. Μιλάμε και για το ζήτημα του ορίου για την πρόθεση μομφής, κατά πόσο θα το χαμηλώσουμε. Ε, σε κάποιες ε, τροπολογίες εκφράζεται η ανησυχία ότι αν μειωθεί το όριο αυτό, θα δημιουργηθούν προβλήματα στην ε, Κομισιόν. Μπορεί να αυξηθούν ε, οι διαφορές μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιόν και να καταλήξουμε σε πολιτική εκμετάλλευση της ε, πρότασης μομφής. Αλλά τα δύο τρίτα που έχουν προβλεφθεί αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δεν επιτυγχάνονται ποτέ. Ίσως θα μπορέσουμε λοιπόν να βρούμε κάποιο συμβιβασμό μεταξύ του να κρατήσουμε το status quo ή να χαμηλώσουμε το όριο υπερβολικά ή πολύ επικίνδυνα. Οπότε... Όπω είπα, θα πρέπει να βρούμε μια συμβιβαστική λύση. Δεν είναι κάτι που θα αποφασίσουμε τώρα, απλά γίνεται μια σύσταση να προσπαθήσουμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ ε, στα, κάποια σταθερότητα, ε, αλλά να υπάρχει μια δυνατότητα σε περίπτωση ε, σημαντικής παραβίασης εκ μέρους της Κομισιόν να μπορεί να παρεύει το Κοινοβούλιο. Το δεύτερο ζήτημα για το οποίο πρέπει να επιτύχουμε κάποιο συμβιβασμό αφορά την ατομική ευθύνη των Ευρωπαίων Επιτρόπων. Όσο περισσότερο κυβερνά το εκτελεστικό φυσικά τόσο πιο συλλογική είναι η ευθύνη αλλά εδώ είναι λίγο διφορούμενο το ποιος είναι ο ρόλος των επιτρόπων. Δεν έχουμε ακόμα εφαρμόσει την συνθήκη της Λισαβόνας οπότε οι επίτροποι που προέρχονται ο καθένας από κάθε χώρα θεωρούνται περισσότερο εκπρόσωποι της χώρας τους παρά του κοινοβουλίου. Ελέγχονται περισσότερο από τις χώρες παρά από Οπότε η ευθύνη των ε, επιτρόπων ενώπιον του Κοινοβουλίου η δυνατότητα μιας πρότασης μορφής παραμένει ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε γιατί υπάρχουν διάφορες απόψεις. Τρίτο ζήτημα σημαντικό η δυνατότητα ακρόασης των υψηλών ε, στελεχών τη Κομισιόν. Αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που εκκρεμεί διαφωνίες μεταξύ κάποιων ευρωβουλευτών και της Κομισιόν όσον αφορά την, τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα, αλλά θεωρώ ότι η δυνατότητα το Κοινοβούλιο να πραγματοποιεί ακρόση των υψηλόβαθμων αξιωματούχων ε, σε, υπαλλήλων σε περίπτωση προβλημάτων με τη συμπεριφορά όχι μόνο των επιτρόπων αλλά και ορισμένων υψηλόβαθμων υπαλλήλων όσον αφορά τις ευθύνες τους και η δυνατότητα να τους υποβάλουμε ερωτήσει όσον αφορά τα καθήκοντά τους είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, χωρίς να επικεντρωθούμε στο σημερινό ζήτημα, που όπως ξέρετε δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Το τέταρτο ζήτημα είναι το ζήτημα της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκεί εξεπλάγει διότι υπάρχουν τροπολογίες κατά του δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και μου έκαναν έκπληξη. Το λιγότερο μπορώ να πω. Και εκεί πιστεύω θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κάποιες συμβιβαστικές λύσεις, διότι έτσι όπως χρησιμοποιείται η νομοθετική πρωτοβουλία στα εθνικά αλλά και στα περιφερειακά κοινοβούλια, καμιά φορά δημιουργεί ανησυχίε, διότι είναι πολλές οι ατομικές πρωτοβουλίες των βουλευτών και που δημιουργούν απλά ε, κορεσμό στις επιτροπές ε, και δεν καταλήγουν ποτέ πουθενά. Αλλά το να υπάρχει ένα οργανωμένο ε, δικαίωμα πρωτοβουλίας από ομάδες οργανωμένες βουλευτών, κάτι δομημένο δηλαδή, όχι να γεμίσουμε με, με πάρα πολλές πρωτοβουλίες το κοινοβούλιο, αλλά να υπάρχει δυνατότητα να αναλάβει μια πρωτοβουλία του κοινοβούλιο μετά, μετά από κάποια έκθεση πρωτοβουλία, α πούμε, να μπορεί να προτείνει κάποιο κείμενο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να βρούμε κάποια συμβαστική λύση που να λαμβάνει υπόψη αυτή την τύχη που θεωρώ είναι σημαντική Παρά ότι δεν σχετίζεται άμεσα με τον πολιτικό έλεγχο της Κομισιόν επί της Κομισιόν ε, ούτως ή άλλως εξακολουθούμε να μιλάμε και για τροποποίηση της συνθήκης. Ε, Μιλάμε για μια πολιτική θέση ουσιαστικά που θα υλοποιηθεί πραγματικά μόνο εφόσον ε, τροποποιηθεί η συνθήκη. Αυτή τη στιγμή ακόμα συζητάμε το μέλλον της Ευρώπης. Όλες μας οι εκθέσεις λοιπόν και αυτή που θα συζητήσουμε αργότερα για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς ε, του συναδέλφου. Όλες αυτές οι εκθέσεις ε, συμπληρώνουν τη δική μας ανάλυση για το μέλλον της Ευρώπης και για τις αλλαγές που θα πρέπει να επιφέρουμε ακόμα και σε επίπεδο συνθήκων αν χρειαστεί για την καλύτερη λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Όπως βλέπετε λοιπόν υπάρχουν πολλά προσυζήτηση Ευχαριστώ όλους τους σκιώδες που παρότι δεν βρίσκονται εδώ αυτή τη στιγμή έκαναν σκληρή δουλειά για τις διάφορες προτάσεις. Θα συνεργαστούμε με όλους τους σκιώδες για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε μια έκθεση όσο το δυνατόν, που την χάνει όσο το δυνατόν ευρύτερη συνένεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μερσέντες. Εξαιρετική παρουσίαση. Σκιώδης. αποουσιάζει ο Έλμαρ Μπρόκ. Ποιος θα μιλήσει από το Ελκό, Γιώργη Σέπφλη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι η φωνή του Έλμαρ Μπρόκ. Ε, μια μικρή δυσκολία. Είναι αδύνατον να γίνω Έλμαρ Μπρόκ. Μια όμως που απουσιάζει, θα ήθελα να ευχαριστήσει την κυρία Μπρέσο για αυτή την πολύ επίκαιρη έκθεση για τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας. Είναι μία από τις κύριες αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου και καθώς έρχεται στο τέλος της η κοινοβουλευτική μας αθητεία είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια αξιολόγηση της κατάστασης σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του επικεφαλής ψηφοδελτίου. Οι αλλαγές που επέφερε η συνθήκη της Λισαβόνας έχουν αλλάξει ουσιαστικά τη σχέση μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διαδικασία εκλογής ε, του Προέδρου της Επιτροπής είναι ένας από τους πυλώνες ε, νομιμότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη και είναι κέρια σημασίας να επικαιροποιηθεί η σταγματική διαδικασία μετά το 2014, όταν ο Ζαν ήταν ο υποψήφιο για την Προεδρία της Επιτροπή από το Συμβούλιο μετά από διαβούλευση με το Κοινοβούλιο. Πρώτα, ε, σε επίπεδο Κοινοβουλίου, οι πολιτικές ομάδες εσωτερικά εξέλεξαν ή υποψήφοι ο οποίο θα μπορούσε να λάβει πλειοψηφία και μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, εγκρίνει την ε, απόφαση αυτή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δημοκρατία. Μόνο ένας υποψήφιος θα έχει την δυνατότητα να γίνει αποδεκτός ε, κατόπιν ε, απόφασης από το Κοινοβούλιο και προεκλογικής εκστρατείας. Ο λαός θα ψηφίσει του χρόνου. Έχω υποβάλει μία τροπολογία η οποία αφορά τη διατύπωση και αναμένω τις προτάσεις ε, των συναδέλφων για αυτό το θέμα και για άλλα θέματα και προσβλέπω σε ε, επικοδομητικές ε, ανταλλαγές απόψεων. Ευχαριστώ Έλμαρ και Γιώργη. Από τους εταιρητικούς και μεταρρυθμιστές δεν βλέπω κανέναν. Φιλελεύθεροι απόντες, Γκουε, Επίσης, οι πράσινοι και αυτοί απουσιάζουν, οι ευθυντοί, το αυτόν και η ΕΝΕΦ. Ο Γιολά είναι τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Όπως βλέπουμε, και οι δύο πολιτικές ομάδες, το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστέ και οι Δημοκράτες, είναι η ραχοκοκαλιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλέπω ότι οι υπόλοιποι απουσιάζουν, δεν συμμετέχουν. Και ελπίζω στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία αυτές οι δύο ομάδες να συνεισφέρουν όπως τώρα στην καλή λειτουργία του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ την Mercedes Presso για αυτή την εξαιρετική έκθεση. Την ε, τελευταία φορά το είπα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει περισσότερα δικαιώματα ε, κοινοβουλευτικού ελέγχου από ότι συνάδελφοι στα εθνικά κοινοβούλια όπου η κατάσταση διαφέρει. Η εκτελεστική εξουσία ελέγχεται με σε διαφορετικό επίπεδο από τα εθνικά κοινοβούλια. Όμως δεν έχουμε λάβει όσα ε, θα έπρεπε. Θα επικεντρωθώ σε δύο-τρία σημεία. Δυσπιστή απέναντι στην εκτελεστική εξουσία. Αυτό είναι ένα δικαίωμα που έχουν τα κοινοβούλια για πρόταση μομφής, για να αποπέμψουν την κυβέρνηση όταν εκείνοι θεωρούν ότι έχει κάνει λάθη. Όπως και με την κυρία Κρεσό, σε περίπτωση που κατηγορηθούν επίτροποι για ε, κάποια πράξη, τότε μπορεί όλο το Σώμα των Επιτρόπων να παρετηθεί. Γι' αυτό νομίζω πως θα έπρεπε να ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για να εξετάσουμε το θέμα της πρότασης μομφής εναντίον μεμονωμένων επιτρόπων. Γνωρίζουμε βέβαια πώς είναι η κατάσταση. Υπάρχει αρνητικό κλίμα που μπορεί να εκτροχιαστεί πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει, χρειάζεται προσοχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση δομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει καθήκοντα για διάστημα πέντε ετών ανεμπόδιστη μπορεί να καταρτήσει και να εκτελέσει το πρόγραμμά της. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να μην έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη των υπολείπων και χρειάζεται λοιπόν να ξεπεράσουμε αυτά τα πολιτικά παιχνίδια και να επικεντρωθούμε στα ουσιώδη. Ο ρόλος των ε, περιφερειών που έχουν νομοθετικές αρμοδιότητες, δηλαδή τα ομόσπονδα κρατήδια στην ε, Γερμανία, ας πούμε, έρχονται σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και τα ομόσπονδα κρατήδια στην ε, Γερμανία εκπροσωπούνται στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο σε διάφορα θέματα, σε θέματα παιδείας ας πούμε κτλ. Υπάρχει εκπροσώπηση λοιπόν σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αυτό θα ήταν ίσως μια καλή λύση, ε, διότι με αυτόν τον τρόπο θα υπήρχε εκπροσώπηση σε τέτοιο επίπεδο. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί επίσης και ένας ειδικό διάβλος επικοινωνίας θεσμικός με, την ευρωπαϊκή, ε, με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ας πούμε όταν έρχεται ο Πρωθυπουργό της Βαυαρία ή της ε, Βορειας Βεσφαλία ε, Βεσφαλίας ε, μπορεί να έρχεται σε επαφή με έναν επίτροπο και να συζητά θέματα περιφερειακής πολιτικής ή θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις δύο πλευρές χωρίς να έχει την ίδια πρόσβαση με εκπροσωπούς της κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα ήταν μια καλή λύση. Τρίτον, οι πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Εδώ υπάρχουν 2.500 τέτοιες πράξεις κάθε χρόνο που έχουν νομοθετικό χαρακτήρα. Στην έκθεσή μου σχετικά με τη διαφάνεια ασχολούμαι με το πόσο μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη αυτών των ε, πράξεων κατ' εξουσιοδότηση, πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία επιτροπολογίας και των άλλων επιτροπών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που συμμετέχουν στη διαδικασία έκδοσης μιας τέτοιας πράξης. Αυτό είναι ένα τομέα στον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε να έχει περισσότερη και καλύτερη πρόσβαση Δυστυχώς πρέπει να αποχωρήσω διότι ψηφίζω στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και λυπάμαι γι' αυτό, αλλά θα ήθελα τέλος να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Ευχαριστώ, Γιώ. Ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη Μερσέντες που μας έδωσε τροφή για σκέψη με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Να σταθώ και εγώ σε τρία σημεία Πρώτον για την νομοθετική πρωτοβουλία. Πολύ συχνά λέγεται πως ε, δεν έχουμε αυτήν την ικανότητα, ε, όπως λέμε ο κύριος Μέσσερ Σμιτ, ε, σε αντίθεση με όλα τα κοινοβούλια του κόσμου. Αυτό δεν ισχύει. Πολλά κοινοβούλια έχουν νομοθετικές αρμοδιότητες και νομοθετική πρωτοβουλία. Είναι πολύ σπάνιο βέβαια να εγκρίνεται νομοθεσία που δεν έχει προταθεί από την κυβέρνηση. Και εσείς κύριε Πρόεδρε το γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι στο Σύνταγμα της ε, Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας θα πρέπει η νομοθεσία να προτείνεται πρώτα από την κυβέρνηση. Είναι βέβαια μια λίγο διαφορετική διαδικασία και αρκετά περίπλοκη. Αλλά στη χώρα μου οποιοδήποτε βουλευτή ε, τη Βουλή των Κοινοτήτων έχει το δικαίωμα νομοθετική πρωτοβουλία και είναι πολύ ε, σπάνιο βέβαια αυτό να οδηγήσει σε νόμο που θα ψηφιστεί από την κυβέρνηση. Υπάρχει όμως αυτό το δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρώτον η Κομισιόν έχει το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας, αλλά έχουμε και εμείς το δικαίωμα να ζητήσουμε από την Κομισιόν να νομοθετήσει, να προτείνει νομοθεσία. Δεν θυμάμαι ακριβώ πόσε τέτοιες περιπτώσεις ε, έχουν υπάρξει στο παρελθόν βέβαια. Όμως υπάρχει αυτή η δυνατότητα η οποία θα μπορούσε να βελτιωθεί. Και νομίζω πως πρέπει να αντικρούσουμε αυτές τις φωνές που λένε ότι όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας. Όχι, στην πράξη έχουμε και επιρροή και τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία νομοθετικής πρωτοβουλίας. Αν όμως αποκτήσουμε και επίσημα το δικαίωμα να ε, προτείνουμε άμεσα και χωρίς παρέμβαση της ε, Κομισιόν, χωρίς να τους το ζητήσουμε ε, ένα νομοθέτημα, τότε θα έπρεπε και ο άλλος κλάδος ε, της νομοθετικής εξουσίας, το Συμβούλιο δηλαδή, να έχει και αυτό ε, το δικαίωμα τούτο. Αυτό το σκεπτικό ότι το, η πρώτη μορφή, το προσχέδιο ενός νομοθετήματος θα πρέπει να προέρχεται από την ε, Κομισιόν, η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Ένωσης και μπορεί ας πούμε να ενώσει τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και τις ε, φωνές όλες, ε, έχει ένα λόγο ύπαρξης. Έχει αποδείξει την αξία του. Αυτή είναι η κοινοτική μέθοδος ε, που λέγαν στο παρελθόν. Αν λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκτήσει επίσημα το δικαίωμα να εισαγάγει νομοθεσία, αυτό θα αλλάξει τα πράγματα. Έπειτα, η πλειοψηφία δύο τρίτων για να απορριφθεί μια πρόταση της Επιτροπής για να αποπεμφθεί αυτή η πρόταση. Υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό μπορεί να ε, γίνει και στα εθνικά κοινοβούλια, όμως αυτό δεν απαιτεί ειδική πλειοψηφία, αλλά απλή πλειοψηφία. Στις περισσότερες περιπτώσεις η εκτελεστική εξουσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει ε, πρόορη διάλυση του Κοινοβουλίου και να προχωρήσει σε εκλογές. Όπως για παράδειγμα και στην Τέταρτη Γαλλική Δημοκρατία, θυμάστε και εσείς κύριε Πρόεδρε. Αυτή η ισορροπία των εξουσιών είναι πολύ λεπτή και νομίζω πως ε, είναι και λίγο επικίνδυνο. Φανταστείτε, ας πούμε, αν προκυρήσονταν προώρες ευρωεκλογέ πώς θα ανατρέπονταν αυτές οι ισορροπίες. Ναι, σίγουρα πρέπει να ελέγχεται η εκτελεστική εξουσία, όμως δεν τόσο απλά τα πράγματα. Χρειάζεται αυτή η δική πλειοψηφία των δύο τρίτων. Δεν είναι άσχημη συμβαστική λύση. Εντάξει, τα δύο τρίτα σας φαίνονται μεγάλο ποσοστό, τα τρία πέμπτα ίσως είναι καλύτερα, μπορεί να είναι η απόλυτη πλειοψηφία ή οποιαδήποτε άλλη μορφή. Εγώ δεν θεωρώ όμως πως αυτή η ισορροπία δεν είναι υγιής. Έπειτα το δικαίωμα μομφής των ε, μεμονωμένων επιτρόπων. Αν δώσουμε στο Κοινοβούλιο την δυνατότητα να αποπέμψει άμεσα έναν επίτροπο, δεν υπομονωμεύουμε την ίδια την ε, θέση του επιτρόπου και η εκτελεστική εξουσία στο σύνολό της είναι υπόλογη και μπορεί να αποπεμφθεί όχι με μονομένα άτομα αυτής. Υπάρχουν, όπως σας είπα, πολύ λεπτές ε, ισορροπίες στο θεσμικό σύστημα της Ένωσης και δεν νομίζω πως είναι κατανάγκη σωστό να, δίνουμε στο να δώσουμε στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να ε, αποπέμψει έναν μεμονωμένο επίτροπο. Υπάρχουν βέβαια οι, οι διοργανικές ε, συμφωνίες ε, και μέσω αυτών μπορούμε να ζητήσουμε από τον πρόεδρο της ε, Κομισιόν να ε, αποπέμψει έναν επίτροπο. Αυτό είναι καινούργια αρμοδιότητα μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Όταν, ας πούμε, σε άλλη περίπτωση δεν μας αρέσει το έργο ενός επιτρόπου, μπορούμε να ζητήσουμε από τον πρόεδρο της Κομισιόν να κάνει κάτι. Και εμέσως, εάν ο πρόεδρος της Κομισιόν δεν το κάνει αυτό, θα πρέπει να ε, λογοδοτήσει στο Κοινοβούλιο με μορφή έκθεσης και μετά εμείς μπορούμε να ασκήσουμε πρόταση μομφής εναντίον ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πρόσφατα δημιουργήθηκε ένας τρόπος που τον οποίο το Κοινοβούλιο έχει πλέον τη δυνατότητα να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για το έργο ενός συγκεκριμένου επιτρόπου, διατηρώντας όμως ε, την εμπιστοσύνη του στο σύνολο του σώματος των επιτρόπων. Κοιτάξτε, εγώ δεν θεωρώ πως πρέπει να φτάσουμε τόσο μακριά και να το τραβήξουμε τόσο πολύ ώστε να απαιτήσουμε να έχουμε το δικαίωμα αποπομπής ενός μόνο επιτρόπου. Ευχαριστώ, Ρίτσαρτ. Να πω κι εγώ δύο λόγια. Πριν προτείνω να κλείσει η Μερσέντε στην τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Συμφωνώ πολύ με όλα αυτά που είπατε. Ιδιαίτερα ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ. Αν παρελπίδα ε, ευοδοθεί το Brexit, παρελπίδα λέω και το απέφχομαι, ε, θα ζητήσω από τον Ρίτσαρτ να αλλάξει η υπηκότητα, να πάρει βελγικό διαβατήριο ή θα προτείνω ψηφοφορία στην Ολομέλεια για να κηρυχθεί Ευρωπαίος πολίτης. Δεν είναι δυνατόν να το χάσουμε. Πάντα θα τον έχουμε ανάγκη τα φώτα του. Ε, συμφωνώ απολύτως για την ε, κοινοβουλευτική πρωτοβούλια. Αυτό ε, στα κοινοβούλια που υπάρχει νομοθετική πρωτοβουλία είναι τελείως θεωρητικό. Ανέφερε στη Γαλλία. Είναι αρκετά ε, κομικό αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία. Ορίζει πάρα πολύ το Σύνταγμα. Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων δαπανών, νέων φόρων, ε, ούτε ε, στο να καθορίζουν νέα αδικήματα ή ποινές για τα αδικήματα αυτά. Την περασμένη εβδομάδα εγκρίθηκε ένα κείμενο μετά από νομοθετική πρωτοβουλία ε, στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση σχετικά με την απαγόρευση, αυτό που ονομάζουμε ε, ε σωματική τιμωρία των παιδιών, ε, το ξύλο που τρώνε από τους γονείς δηλαδή, και απαγορεύεται στους γονείς να δέρνουν τα παιδιά τους ή να τους ε, υποβάλλουν σε ψυχολογική πίεση ακόμα και να τους βάζουν τις φωνές. Αυτό το ψήφισαν ε, κατά πλειοψηφία άνθρωποι που δεν έχουν γεννήσει φαίνεται παιδιά στη ζωή τους, αλλά από νομικής πλευράς δεν προβλέπει καμία ποινή αυτό. Άρα αυτόματα θα ακυρωθεί από το ε, Συνταγματικό Συμβούλιο, γιατί και σωστά το Συνταγματικό Συμβούλιο ορίζει ότι ε, όταν ένας νόμος παραβιάζεται και δεν προβλέπεται ποινή για αυτόν, για αυτή την παράβαση του νόμου, τότε δεν είναι νόμος. Ε, και σχεδόν όλα τα νομοθετικά καθεστώτα ε, βλέπουν να καθορίζει τη μερίσια διάταξή τους από κυβερνήσεις. Ή από την άλλη βέβαια μπορεί να έρθει νομοθετική πρωτοβουλία από το Κοινοβούλιο, αλλά με την συμφωνία του, κοινοβου... του της ή ε, της κυβέρνησης, δηλαδή κάποιοι βουλευτές της συμπολίτευση να το προτείνουν. Και όπως είπε και ο Ρίτσαρτ, ουσιαστικά ε, μέσω των ψηφισμάτων που εμείς εγκρίνουμε σε κάθε ολομέλεια, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει κάποια δράση σε κάποιο τομέα. Άρα, ε, ξέρω εγώ, ζητούμε να τροποποιηθούν κάποιοι κανονισμοί και κατά αυτόν τον τρόπο είναι ένα είδος νομοθετικής πρωτοβουλίας. Ε, σε κάθε νέα ε, θητεία κάνουμε διοργανική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορούμε την επόμενη φορά να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και να καταστήσουμε πιο δεσμευτική πολιτικά μια τέτοια διάταξη ε, στη συμφωνία που θα συνάψουν ε, οι επόμενοι βουλευτές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ταυτόχρονα συμφωνώ με τον Ρίτσαρτ σε αυτό που ε, είπε να διατηρηθεί ο συλλογικό χαρακτήρα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως γίνεται και με τις κυβερνήσει. Πρόταση μορφή κατά μεμονωμένου επιτρόπου σίγουρα όχι. Δεν ε, μπορούμε να εφεύρουμε διαδικασία καθαίρεση, σαν σκότω στην πεθερά του ένα επίτροπο, α πούμε ή ε, έκλεψε λεφτά από τα Ταμεία Συνοχής αλλά σε μια τέτοια περίπτωση αυτό είναι θέμα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκείνος θα πρέπει να λάβει πρωτοβουλία. Μπορούμε να το αναφέρουμε και αυτό στην διοργανική συμφωνία που θα υπογράψουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά χρειάζεται προσοχή να μην αμφισβητήσουμε το συλλογικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσθέτω ότι το πρόβλημα το είδαμε το 1999 στην Επιτροπή Σαντέρ τότε, όταν αποκαλύφθηκε ότι δύο επίτροποι είχαν παραβιάσει την κοινοτική ε, νομοθεσία και τον κώδικα δεοντολογίας. Και ο πρόεδρος Σαντέρ θα μπορούσε να τους είχε ξεφορτωθεί, αλλά θεώρησε ότι είναι συλλογική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό έλεγε τότε και το Κοινοβούλιο. Κάτι λέει ο κύριο Κόρμπετ εκτός ε, μικροφώνου. Α, δεν είχε το δικαίωμα ο Σαντέρ να τους διώξει. ωραία. Ε, τότε παρετήθηκε λοιπόν όλη η Επιτροπή Σύσσωμη υπό την απειλή της ε, πρότασης στο Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά τη μομφή και τη δυσπιστία, Ρίτσαρτ, στις δικές μας δημοκρατίες είχαμε πολλές εμπειρίες που κατέληξαν ε, στην κατάλυση της δημοκρατίας και την εξαφάνισή της. Ή σε καταχρήσεις. Στη Γαλλία γινόταν αυτό στην τέταρτη γαλλική δημοκρατία, όπου προβλέπεται από το Σύνταγμα ότι για να ρίξεις κυβέρνηση χρειάζεται ειδική πλειοψηφία στη Βουλή. Τύπου 2 τρίτων, δεν θυμάμαι απόλυτη πλειοψηφία, κάτι τέτοιο, στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Αλλά στην πράξη τι γινόταν. Πολύ συχνά είχαμε προτάσεις μορφής και αρκούσε απλή πλειοψηφία έτσι ώστε πολιτικά η κυβέρνηση που δεν ήταν βέβαια νομικά υποχρεωμένη να παραιτηθεί, να οδηγεί το στην παρέτηση. Αν δεν υπάρχει λοιπόν κάποια ασφαλιστική δικλίδα εδώ, είτε το δικαίωμα διάλυσης της Βουλής, όπως ανέφερε ο Ρίτσαρτ, ή κάτι άλλο που λέει το Γερμανικό Σύνταγμα, δυνατότητα πρότασης μορφής, αλλά μόνο σε περίπτωση που νέα ε, πλειοψηφία αντικαθιστά την κυβέρνηση που καθερεί. Δηλαδή είναι ένα είδος επικοδομητικής πρότασης μορφής. Εδώ ε, αυτά κινδυνεύουν να έχουν κάποια προβλήματα και συνιστώ και εδώ πρόσοχη. Αυτά, Μερσέντες, παρακαλώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη γιατί βλέπω ότι έχουμε καθυστερήσει και με τις άλλες εκθέσεις. Όπως είχα πει, ε, η συζήτηση κατέληξε σε τρία-τέσσερα σημεία για τα οποία έχουμε και τις περισσότερες τροπολογίες ε, και με τους κοιόδης η συνεργασία μας θα εστιαστεί σε αυτά. Όσον αφορά την ομοθετική πρωτοβουλία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλοι μας οι συνομιλητές, οι εξωτερικοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα διάφορα ε, προευρωπαϊκά κινήματα θεωρούν ότι αποτελεί σοβαρό περιορισμό των εξουσιών του Κοινοβουλίου αυτό το θέμα είναι προφανές και εγώ συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν ότι συχνά δεν χρησιμοποιείται σωστά στα Εθνικά Κοινοβούλια. Δηλαδή όταν γίνεται κατάχρηση ένα σωρό νομοθετήματα παραμένουν στα σιρτάρι. Και σπάνια, πολύ σπάνια καταλήγουν σε κείμενα αφού η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει για να τα βάλει σε τάξη. Τώρα, ε, το δικό μας κοινοβουλίο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ε, ε, έχει πολύ τεχνικό προσωπικό και δυνατότητες για πολλές τροπολογίες στις περισσότερες χώρες τα κείμενα βασίζονται στα, στις επιθυμίες των κυβερνήσεων ενώ εδώ οι τροπολογίες μπορεί να είναι πολύ σημαντικές και να γίνουν μεγάλες αλλαγές οπότε υπάρχουν και μεγάλες τεχνικές δυνατότητες παρέμβασεων τώρα όπως είπα μπορούσαμε, θα μπορούσαμε να το σχετίσουμε με την έκθεση πρωτοβουλίας που εγκρίνονται από τη διασκέψη των Προέδρων σε περιορισμένο αριθμό. Κάθε επιτροπή διαθέτει συγκεκριμένο αριθμό. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι τροποποιώντας τις ε, συνθήκες ε, μετά από μία έκθεση πρωτοβουλίας θα μπορούσαμε να αλλάξουμε λίγο την υπάρξουσα νομοθεσία. Αυτό είναι το πιο πιθανό ή θα μπορούσαμε να έχουμε ένα νομοθετικό κείμενο. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα το κάνουν ατομικά οι βουλευτέ. Θα υπάρξει μια κοινοβουλευτική διαδικασία ολόκληρου του Κοινοβουλίου για να οδηγηθούμε σε κάποια πρωτοβουλία. σω θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό ώστε να αποφύγουμε τι καταχρήσει και να αποφύγουμε να υποβαθμιστεί και η ποιότητα τη νομοθετική ε, ε, πρόταση του Κοινοβουλίου αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τους επιτρόπους, όλοι βασιζόμαστε ε, στην υπόθεση ότι η Κομισιόν είναι πιο πολιτική, ότι η διαδικασία των κορυφαίων εκπρόσωπων των Spitzenkandidat θα συνεχίσει. Αλλά αυτό, ξέρετε, δεν είναι βέβαιο, διότι πολλά κράτη είναι κατά. Η περίπτωση λοιπόν η Κομισιόν να έχει διαφορετική σύνθεση, ενδεχομένως και με επιτρόπους ε, που εναντιώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που θα υιοθετούν στάσεις κατά των συνθήκων, είναι ένα σενάριο που δεν αποκλείεται. Α σκεφτούμε λοιπόν, να έχουμε υπόψη μα ότι μπορεί να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ε, με περιορισμού φυσικά όσον αφορά την επιχειρηματολογία. μπορεί εκεί να υπάρξει περισσότερος έλεγχος από το Κοινοβούλιο όσον αφορά κάποιου επιτρόπους με μια συγκεκριμένη πράξη. Τώρα όσον αφορά το όριο, Συμφωνώ, δεν μπορούμε να το μειώσουμε υπερβολικά. Αλλά μπορούμε να φανταστούμε κάποιο ποσοστό το οποίο ταυτόχρονα θα διασφαλίζει ότι θα είναι δυνατό να υπάρξει μια συμφωνία χωρίς να απαιτείται υπερβολικά ευρεία συμφωνία η οποία δεν είναι εφικτή. Δεν συζητήσαμε για το κατακόρυφο χαρακτήρα του ελέγχου των κοινοβουλίων που σχετίζονται με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών. Ένα πρόβλημα δεν είναι το κατά πόσο μπορούν να συναντήσουν τους επιτρόπους στα Εθνικά Κοινοβούλια. Το ζήτημα είναι όσον αφορά την συχνά άμεση εφαρμογή από τα περιφερειακά κοινοβούλια των ευρωπαϊκών οδηγιών. Τι γνωρίζουμε εμείς, πώς ελέγχουμε δηλαδή την εκτέλεση που είναι απαραίτητα πολύ επίπεδη. Διότι Υπάρχουν τα κράτη και μερικές φορές αντικαθίστανται αυτά ή συμπληρώνονται από τα περιφερειακά κοινοβούλια. Συχνά δεν γνωρίζουμε καθόλου τι συμβαίνει εκεί. Σιγά σιγά με τις διάφορες κοινοβουλευτικές ε, συνελεύσεις ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και βουλευτές ε, των κρατών μελών καταφέρνουμε πάλι να συντονιστούμε κάπως. Ε, καταφέρουμε να συντονιστούμε όμως με τα περιφερειακά κοινοβούλια καθόλου. Δεν έχουμε καμία σχέση και ότι αυτοί εκτελούν, εφαρμόζουν μερικές φορές καλά, άλλες φορές άσχημα, άλλες φορές πολύ άσχημα τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Είναι πρόβλημα συντονισμού. Το οποίο μπορούμε να υπογραμμίσουμε, αλλά φυσικά απαιτείται να κάνουμε κάτι νομοθετικά ε, ε, ρυθμιστικά ε, με κάποιες συμφωνίες διοργανικές ή με κάποιο άλλο μέσο το οποίο θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Θα το ξανασυζητήσουμε αφού ολοκληρωθεί η μελέτη των συμβιβαστικών τροπολογιών. Ευχαριστούμε κυρία Μησηγήτρια. Πώς θα έχει τώρα η συνέχεια και το χρονοδιάγραμμα για την έκθεσή σας. Εδώ στην Επιτροπή μας θα ψηφίσουμε στις 22 Ιανουαρίου και στην Ολομέλεια πάει το Φεβρουάριο. Λοιπόν, θα σας προτείνω τώρα να περάσουμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης, που είναι η εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Το λόγο έχει η Μαϊτέ Παγάσα Ορτουντούα, που είναι και η αρμόδια εισηγήτρια και μόλις κατέφθασε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι μήνες τώρα ολόκληρους Oui. Vale. Ε, έλεγα λοιπόν ότι εδώ και μήνες ολόκληρους εργαζόμαστε ε, για το θέμα αυτό. Και ε, έχουμε πολλές ελπίδες ε, για το συγκεκριμένο θέμα. Παρακαλώ, επειδή δεν έχουμε χρόνο, τις οπολογίες να τις καταθέσετε μόνο στα αγγλικά. Ένα από τα βασικά ζητήματα για τα οποία ανησυχούσαμε και ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συνεργασία στην έκθεση αυτή. Ήταν το εξής. Μιλούμε για τη δημιουργία μιας πολιτικής κοινότητας όταν αναγνωρίζουμε την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Αλλά δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί πλήρως αυτή η δυνατότητα και δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο υπάρχουν ταυτότητες αποκλειόμενες και αποκλειστικές που σηκώνουν κεφάλι στην ε, ε, Ευρώπη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον να εργαστούμε σε αυτό το θέμα μέχρι που καταφέραμε να το εφαρμόσουμε αυτό και να το υλοποιήσουμε στην πράξη. Γιατί δεν μπορεί να είναι ένα διάχυτο τέτοιο ε, σώμα που δεν έχει καμία μορφή και καμία Ισχύει. Έχουμε περιορισμούς στην έκθεση και ε, χώρου, γι' αυτό δεν τα έχω γράψει όσα ήθελα να γράψω, θα κάνω και τροπολογίες. Η έκθεση έχει ως στόχο να είναι όσο γίνεται πιο κατανοητή και εύληπτη. Είδαμε τα διάφορα δικαιώματα που ορίζονται από τις συνθήκες και φυσικά αρχίσαμε από τα πολιτικά δικαιώματα. Το θέμα της ενεργής συμμετοχής υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ζουν εκεί που γεννήθηκαν και που έχουν δυσκολία ε, στη συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθε της χώρας που ζουν. Και αυτό είναι πραγματικά ακόμα μια πραγματικότητα που δεν αφήνει τους πολίτες να εκφραστούν. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει κάτι τέτοιο ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τονίζουμε στο κείμενό μας αυτό. Επίσης, ε, σκεφτήκαμε πώς μπορούμε να καταργήσουμε όλα αυτά τα εμπόδια πέρα από τα κράτη-μέλη. θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες δομές που υπάρχουν ή που δεν υπάρχουν. Αν υπάρχουν τόσο το καλύτερο, ε, γιατί είναι πιο αποτελεσματικό, για να έχουμε ένα ε, ρόλο διαμεσολαβητικό, για να καταργηθούν και να αρθούν κάποια εμπόδια όταν δεν είναι απόλυτα και να είναι καλύτερη η συμμετοχή πολιτική, κοινωνική των πολιτών. Για τους πολίτες που δεν ζουν, επαναλαμβάνω, στον τόπο που γεννήθηκαν. Αυτές οι δομές λοιπόν διαμεσολάβησης θεωρούμε ότι μπορεί να είναι σημαντικές και θα μπορέσουμε να τις συζητήσουμε κιόλας. Για την ελεύθερη κυκλοφορία. Είναι μεν από τα δικαιώματα που καταλαβαίνουν από ένστικτο καλύτερα οι πολίτες, αλλά όταν προσπαθούμε να την εφαρμόσουμε στην πράξη αυτή την ελεύθερη κυκλοφορία, ερχόμαστε αντιμέτωποι με εμπόδια και μάλιστα με διακρίσεις. Δεν λέω ότι ε, όλες αυτές οι περιπτώσεις διακρίσεων είναι γνωστές και καταγγέλλονται, γιατί πολλές φορές όταν έχει κάποιος πρόβλημα ε, δεν το καταγγέλει. Συμβιβάζεται, Είναι κρίμα όμω, γιατί αν δεν καταγγέλλονται αυτά τα πράγματα, δεν μπορούν να γίνουν οι απαραίτητε νομικέ προσαρμογέ και να βελτιώνεται η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είναι κάτι που έχει βγει στο προσκήνιο, γιατί στις διαπραγματεύσεις ε, για τον Brexit ε, ακριβώς κυριαρχούν αυτά τα θέματα των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν σε διαφορετική χώρα από την πατρίδα τους. Επίσης, μιλήσαμε και για το θέμα της προξενικής προστασίας. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα, ιδιαίτερα σε έκτακτες περιστάσεις και σε κρίσεις για πολίτες που βρίσκονται σε τρίτες χώρες. Η προξενική προστασία είναι πολύ σημαντική και μπορεί να ασκείται με τρόπο αλληλέγγυο, δηλαδή μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Δεν είναι γνωστό αυτό το δικαίωμα, παρότι πολύ σημαντικό ο κόσμος δεν το γνωρίζει πολύ. Πρέπει να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να γίνει πολύ πιο γνωστό και ιδιαίτερα σε έκτακτες περιστάσεις και σε πολύ σκληρές καταστάσεις να το ξέρουν οι πολίτες και να το χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους. Υπάρχουν πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και κάποια άλλα που προτείνουμε. Και βέβαια, όλους αυτούς τους μήνες συζητούσαμε με νέους, με μεγαλύτερους σε ηλικία, με ειδικού, με διαμεσολαβητές, με ανθρώπους που εργάζονται σε διάφορες διοικήσεις ή θεσμούς. Και κάτι που γνωρίζουν όλοι και το λέγουν είναι ότι κάτι που λειτουργήσε πάρα πολύ καλά ήταν τα προγράμματα που συνδέονταν με τον έρασμο. Θα πρέπει να ξαναδούμε λοιπόν αυτά τα θέματα των νέων και της εκπαίδευσης. Έχουμε μια, ε, ένα κεφάλαιο στην έκθεση για τις ε, επαγγελματικές διαπιστεύσεις και αναγνωρίσεις, για να μην έχουμε ενεργεία, για να μπορεί ο κόσμος να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εργάζεται. Και αυτό έχει να κάνει με τις αναγνωρίσεις των πτυχίων και τις ισοτιμίες των πτυχίων. Εκεί χωράει πολύ μεγάλη βελτίωση. για να μπορούν οι νέοι μας να βιώνουν περισσότερο αυτή την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Είναι πολλά τα θέματα, πολύ περισσότερα από αυτά που σας αναφέρω. Θέλω όμως να τονίσω το εξής, έτσι καταλεκτικά. Χωρίς να ζητάμε τον ουρανό μετάστρα, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα απαιτούμε. Έχουμε κάποιες δυνατότητες και μάλιστα νομικές δυνατότητες. Αυτό που θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να κάνουμε είναι να σκεφτούμε να κωδικοποιήσουμε κάπου όλα τα ειδικά δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και τις επιπτώσεις τους και να συντάξουμε ένα είδος καθεστώτος των δικαιωμάτων του πολίτη. Δεν ζητάμε αναθεώρηση της συνθήκης, αξιοποίηση του άρθρου 25 για να ενώσουμε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, από την ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην είναι κατακαιρματισμένες αυτές οι διατάξεις και τα δικαιώματα κάπως αδέσποτα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν τα εντάξουμε όλα σε ένα σώμα, σε ένα κανονισμό, μπορούμε πραγματικά να δημιουργήσουμε ένα τεράστιο δυναμικό, να γίνεται ορατό αυτό, να φαίνεται, να προβάλλεται και να εμπνέει για νέα δικαιώματα και με μια άλλη ματιά και αυτό νόμιμοποιεί και δίνει και πολύ μεγάλη αξιοπιστία στην προσπάθεια που κάνουμε. Τουλάχιστον όσοι θεωρούμε ότι η καλύτερη ευκαιρία μας για το μέλλον είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να συνεργαστώ με όλους, ελπίζω να μην μακρηγόρησα και να μην επεκτάθηκα πάρα πολύ και σας ευχαριστώ και τη Γραμματεία και τους συναδέλφους και τους υπαλλήλους Ευρωπαϊκής Επιτροπής που με βοήθησαν πάρα πολύ στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ κυρία εισηγήτρια. Λοιπόν, σκιώδης, ΕΛΚ. εγωσιάζει ο Μίχαλ Μπόνι. Ο συντονιστής ε, έχει καμία ε, εντολή να πει τίποτα. Όχι, δεν έχω. Αυτή τη στιγμή το ΕΛΚ δεν έχει τίποτα να πει παρά μόνο να ευχαριστήσει τη Μάιτε για τη δουλειά της. Ωραία. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο κύριος Αντιπρόεδρος Σίλβα Περέρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Θα ήθελα να εκφράσω κι εγώ την ε, ευγνωμοσύνη μου στον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά του. Συμπεριέλαβε τις ε, προτάσεις μας ε, και τα σχόλιά μας που είχαμε κάνει στην αρχική ανταλλαγή απόψεων. Θεωρούμε πως η έκθεση αυτή πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση και συμφωνούμε απόλυτα με αυτή τη γενικότερη προσέγγιση που υιοθέτησε ο εισηγητής. Στηρίζουμε επίσης την έμφαση που δόθηκε στα πολιτικά δικαιώματα, στην ελεύθερη κυκλοφορία και την προστασία των καταναλωτών. Ωστόσο, τώρα καιρός είναι να προχωρήσουμε κάποια επιμέρους σημεία λίγο περισσότερο. Χαιρετήσουμε λοιπόν την αναφορά στο θέμα της εκπαίδευσης ε, για την ηθαγένεια, την υπηκότητα. Θεωρούμε πως είναι πολύ καλή η έμφαση που δόθηκε, διότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τι δικαιώματα έχουν και τι σημαίνει το να είναι κανείς Ευρωπαίος ε, πολίτης. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να γίνουν επενδύσεις ε, σε εκστρατείες, ευαισθητοποίησης και ενημέρωση, έτσι ώστε να αυξηθεί η ενημέρωση για την ευρωπαϊκή υπηκότητα. Επίσης, ε, θέματα διάκρισης. Η έκθεση αυτή, όπως βλέπετε, θα πρέπει να είναι ένα μανιφέστο κατά των διακρίσεων. Είτε αυτές οι διακρίσεις αφορούν ε, ρατσισμό, είτε ξενοφοβία, είτε την εθνικότητα, το φύλλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό. Τρίτον, και είναι σημαντικό αυτό που θα πω, η έκθεση αυτή θα ε, δημοσιευθεί λίγο μετά τις ευρωεκλογέ. Θέλουμε λοιπόν ε, να τονίσουμε πως πρέπει να αναγνωριστεί η μεγάλη σημασία των ευρωεκλογών, των συγκεκριμένων ευρωεκλογών. Γι' αυτό λοιπόν ε, ζητούμε να γίνουν επενδύσεις στην διάδοση αυτή ακριβώ της αλήθειας, ε, του πόσο σημαντικές είναι οι εκλογέ, γιατί η ψήφος μπορεί να κάνει τη διαφορά, ακόμα και αν είναι μόνο μία. Το να πάει κανεί στις κάλπες έχει πάντα θετικέ ε, συνέπειες και είναι κάτι που πρέπει να το πάρουμε όλοι στα σοβαρά. Και δεν θα και πως μπορεί αυτό να αλλάξει το πολιτικό τοπίο και τις ε, πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στις ε, ζωές των ανθρώπων. Πρέπει να περάσουμε λοιπόν αυτό το μήνυμα ότι οι ευρωεκλογέ είναι πάρα πολύ σημαντικές και έχουν αντίκτυπο στη ζωή όλων. Ας πάρουμε λοιπόν ιδέες από τα όσα έχουμε ήδη συζητήσει, από τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου, από τη διαδικασία του επικεφαλής ψηφοδελτίου, και να τονίσουμε ότι όλα αυτά προσθέτουν ακόμα περισσότερη αξία στην ευρωπαϊκή διάσταση. Χρειάζεται όμως να εκφράσουμε και τις ανησυχίες μας για τις ενδεχόμενες παρεμβάσεις ή τη χειραγώγηση των ευρωεκλογών, διότι εφόσον αυτό συμβεί, αυτό υπονομεύει την βούληση του εκλογικού σώματος. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να παρέμβει στην εκλογική διαδικασία και να χειραγωγήσει τις εκλογές. Και αυτό σημαίνει ότι παραβιάζονται τα πολιτικά δικαιώματα των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνοψίζοντας λοιπόν, ε, θα ήταν καλό να σταλεί ένα μήνυμα για τη χρηματοδότηση. Να πούμε πως είμαστε κάθετοι σε οποιαδήποτε διαδικασία περικοπών που θα υπονομεύσει τις ε, αξίες μας. και θα συρρυκνώσει τις δυνατότητές μας για ενημέρωση του κοινού σχετικά με, την, ε, με τα πολιτικά του δικαιώματα και τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία. Αλλά θέλουμε να στηρίξουμε την εισηγήτρια, διότι η έκθεση αυτή είναι μια εξαιρετική βάση για μελλοντική εργασία. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Οι υπόλοιπε πολιτικές ομάδες απουσιάζουν. Οπότε θα προτείνω στη Μάιτε να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Θέλω να πω στον συνάδελφο από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες ότι είμαστε πανευτυχείς ε, που συμπίπτουν οι απόψεις μας για το θέμα αυτό και το τι θέλουμε να κάνουμε στην έκθεση. Για λόγους χώρου δεν μπορέσαμε να γράψουμε όλα όσα θέλαμε. Αλλά το θέμα είναι και ένα θέμα σεβασμού ε, προς εσάς. Θέλουμε αυτό το πίνακα να το ζωγραφίσουμε όλοι μαζί. Ε, μια συλλογική προσπάθεια, ένα συλλογικό έργο. Η δική μου πρόταση είχε τη φιλοδοξία να είναι μια καλή βάση, μια αφετηρία για τη συζήτηση που θα βελτιώσει όσο μπορεί την έκθεση. Για ένα θέμα που αυτή τη στιγμή κυριαρχεί και εμφανίζεται ως στρατηγικό γιατί διακυβεύεται το ίδιο το μέλλον μας στην Ευρώπη που είναι η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ κύριε Συγήτρια. Θυμίζω τη συνέχεια, τη χρονική ε, για τις εργασίες μας. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 13 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα και όπως είπε και η συγκεκριά μας παρακαλώ μόνο στα αγγλικά για λόγους χρονικούς. Η ε, ε, συζήτηση για τις τροπολογίες και ψηφοφορία θα γίνει στην Επιτροπή μας στις 22 Ιανουαρίου και η έγκριση ε, θα πάει το Φλεβάρι ή το Μάρτιο στην Ολομέλεια. Οπότε, μπορούμε να περάσουμε τώρα στην έκθεση του Γιώργη Σόεπφλινγκ για την εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινή δήλωσης που ε, εξασφαλίζει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών. Έχεις το λόγο, παρακαλώ, Γιώργη Σεπφλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως θα γνωρίζετε κάποιοι από εσάς, η Επιτροπή μας έχει ήδη συζητήσει αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόβλημα. Συνδυάζεται και με το όλο ζήτημα του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υπόβαθρο έχει ως εξής. Κάθε κυβέρνηση αναθέτει ένα κομμάτι του έργου της σε ειδικευμένους οργανισμούς. Δεν είναι ιδιαιτερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. είναι λίγο δύσκολο να το περιγράψουμε. Υπάρχουν πάνω από 40 οργανισμοί και ε, όργανα παρεμφερεί με οργανισμούς. Έτσι έχει αναπτυχθεί αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικά είναι κοινοπραξίες, ε, κάποια έχουν άλλη χρηματοδότηση, κάποια έχουν 100% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλοι εν μέρη. Είναι περίπλοκη η διάρθρωση και ελπίζω στην εκθέση μου να καταφέρω κάπως να ξεκαθαρίσω τα πρώτα, να τα βάλω λίγο σε τάξη, χωρίς να πω ότι είμαι τέλειος φυσικά. Το σκεπτικό στο οποίο βασίσαμε αυτή την έκθεση είναι το ζήτημα της διακυβέρνησης. Δεν ε, αποτελεί έκθεση επίκριση του έργου των οργανισμών αυτών των επικεντρωμένων. Αναφέρουμε απλά το πρόβλημα της λογοδοσίας και της ε, εποπτείας. Αυτή τη στιγμή οι οργανισμοί, χωρίς να μπορούμε να είμαστε ακριβείς, ε, διότι είναι δυναμική διαδικασία, απασχολούν πάνω από 9.000 ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικός ο προπολογισμό. Το θέμα με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς είναι ότι ε, λειτουργούν ε, αποστασιοποιημένοι από πολιτική παρέμβαση. Αν δείτε τι συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι κεντρικές τράπεζες δεν δέχονται μεγάλη πολιτική παρέμβαση. Οι νομοθέτες λοιπόν δυσκολεύονται να ασκήσουν εποπτεία. Ελάχιστη είναι η πολιτική επιρροή, ε, η οποία αλλού είναι αποδεκτή και αλλού όχι. Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί λειτουργούν κυρίως τεχνοκρατικά, ασχολούνται με πολύ περίπλοκα ζητήματα και εποπτεία όπου υπάρχει γίνεται με νομικά μέσα. αποπολιτικοποιημένα εντελώς και στους περισσότερους τομείς αυτό είναι ε, αποδεκτό, αλλά αλλού τίθενται ερωτηματικά. Όσον αφορά τώρα τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κομμάτια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης παρότι ανεξάρτητη και αυτόνομη και είναι απευθείας υπόλογοι στους ψηφοφόρους. Αυτό προσπαθώ να ε, τεκμηριώσω εδώ στην έκθεση. Κάποιοι από εσάς θα γνωρίζετε το έγγραφο αυτό το οποίο έχει εκπονήσει η Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η καθηγήτρια Λεμβός που ήταν σε ακρόαση εδώ ε, πρόσφατα, ονομάζεται Κοινοβουλευτική Εξέταση, Κοινοβουλευτικό Έλεγχο των Αποκέντρωμένων Οργανισμών. Είναι πολύ καλό έγγραφο. Ουσιαστικά οι οργανισμοί που καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο, αλλά θεσμικά είναι ξεχωριστοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτόνομοι. έχουν θεσπιστεί δυνάμει του άρθρου 352 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2012 υπήρξε μια κοινή δήλωση και προσέγγιση για το τι είναι αυτοί οι οργανισμοί και που βρίσκονται, αλλά δεν υπήρξε διοργανική συμφωνία. Το Κοινοβουλίο έχει το δικαίωμα εξέταση, το περιγράφω λεπτομερό στον αγγραφό, με διάφορου τρόπου. Και στη συνέχεια πραγματοποιώ κάποιε συστάσει στην έκθεσή μου βάσει του έργου των συνεργατών μου και του ευχαριστώ όλους. Εγώ επισκέφθηκα τρεις οργανισμούς, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη Βιέννη, την Τσέπολ, στη Βουδαπέστη και τον Γκαλιλαίο GSA στην Πράγα. Ε, έκανα δηλαδή ένα tour στην Κεντρική Ευρώπη. Τα όσα έμαθα τα θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα και με βοήθησαν πολύ. Οι συστάσεις μου ουσιαστικά είναι ότι μπορούν και πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες απλούστευσης των διατάξεων στους κανονισμούς χρηματοδότησης των οργανισμών όσον αφορά τη διακυβέρνησή τους και την λογοδοσία τους, λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους τύπους των οργανισμών, ομαδοποιώντας τους ε, ανάλογα με τις ειδικεύσεις τους, τα καθηκόντα τους και καθορίζοντας τις γενικές αρχές που διέπουν τη σχέση μεταξύ των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αποκεντρωμένων αυτών οργανισμών ορισμένα από αυτά τα ζητήματα, πιθανότητα και όλα, θα πρέπει να εξεταζονται σε εκτιμήσει αντικτύπου κάθε φορά που προτείνεται ίδρυση ενός οργανισμού. Υπάρχει ένας νέος για τα εργασιακά ζητήματα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα γενοφάσκια και ένα από τα πράγματα που ανακάλυψα και το στο ιστορικό ότι κάθε φορά που υπάρχει κάποιο πρόβλημα λέμε ας ιδρύσουμε έναν οργανισμό υπερβάλλω λίγο, αλλά κάπως ε, έτσι μοιάζει. Ε, ουσιαστικά εγώ κάνω έκκληση να αξιολογήσουμε την υλοποίηση της κοινή προσέγγισης σε όλες τις, τις πτυχές με λεπτομερή αναλυτικά έγγραφα παρόμοια με αυτά που εκπονήθηκαν το 2010 να δούμε με μια νέα ματιά, δεδομένου ότι έχει περάσει κάποιο χρόνος, ε, να δούμε κατά πόσο μπορεί να υπάρχει μια διοργανική συμφωνία για τους οργανισμούς αυτούς. Η συμφωνία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξει που θα αναθεωρούνται κάθε 5 ή 6 χρόνια ε, για τη λειτουργία τους, την ίδρυσή τους, ε, τη σχέση μεταξύ των οργανισμών και των ευρωπαϊκών θεσμών. Το πρόβλημα αυτό είναι κάπως ιδιαίτερο το θα, και θέλω να το σημειώσω. Ε, ο κάθε αποκεντρωμένος οργανισμός έχει ιδιαίτερη σχέση με το κράτος όπου εδρεύει. Είναι κάπου σαν μια ιστορία αγάπης, ε, για να το πω κάπως υπερβολικά. Και το κάθε κράτος μέλος ε, κάνει ό,τι μπορεί για να διακρατήσει τον οργανισμό αυτό στο έδαφος του. Και αυτό σίγουρα είναι μια πτυχή σημαντική όσον αφορά τη λειτουργία κάθε οργανισμού. Στην έκθεση Επίση προτείνουμε το Κοινοβούλιο να πραγματοποιεί ετησίω μια συζήτηση για τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση των αποκεντρωμένων οργανισμών, το οποίο θα προηγείται μια συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μα. Τη οποία θα προηγείται μια συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε χωρί καμία καθυστέρηση. Επίση, προτείνουμε οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί να υπόκεινται στου ίδιου κανόνε, να υποβάλλουν του ίδιου κανόνε διαφάνεια όπω το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και οι ίδιοι κανόνε να ισχύουν για όλους τους ε, ενδιαφερομένους ε, που σχετίζονται με αυτούς τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Συχνά δεν τους γνωρίζουμε, οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί τους γνωρίζουν, αλλά όχι εμείς. Και μετά τίθεται και ένα ζήτημα αλλαγή τη συνθήκη. Προτείνουμε σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγή ε, τη συνθήκη να εξεταστεί το πώ οι συνθήκε μπορούν ειδικότερα όσον αφορά το άρθρο 13 ε, και τα άρθρα 9, 291 και 290 της Σύνθηκης Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλαβα σχόλια από πολλέ επιτροπέ. Άλλε επιτροπέ ε, επιβλέπουν πολλές, ε, πολλούς οργανισμούς. Η ΛΥΜΠΕ νομίζω επιβλέπει εννέα. Εμείς επιβλέπουμε μία, την αρχή των πολιτικών κομμάτων. Αλλά είναι και κάτι καινούριο ουσιαστικά. Αυτό ήθελα να πω στην παρούσα φάση. Ε, θα ήθελα να ε, δω και τα δικά σχόλια που θα καταθέσετε υπό μορφή τροπολογιών. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σιγητά. Οι για τους σοσιαλιστές μεσέδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον συναδελφό Σέπλεν για τις προσπάθειές του και, για την έκθεση, και η έκθεση αυτή από το κέντρο έρευνας ε, που προέρχεται από την πολύ ενδιαφέρουσα ε, καθηγήτρια και η έκθεση αυτή λοιπόν μας έδωσε ένα πλαίσιο μας περιγράφει μια άλλη πτυχή του ελέγχου των εκτελεστικών δραστηριοτήτων που συμπληρώνει πολύ καλά και τις δικές μου προσπάθειες όπως είναι προφανές στους αποκεντρωμένους οργανισμούς εκχωρούμε ένα κομμάτι της εκτελεστικής εξουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συχνά σημαντικές πτυχές. Αναμφίβολα λοιπόν χρειάζεται να μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα τι κάνουν και ενδεχομένως να μπορούμε να επιβάλλουμε και κάποια ανακατεύθυνση, κάποιον επαναπροσανατολισμό. ανατολισμό ε, αυτή η πτυχή της ανεξαρτησίας που είναι εξαιρετικά χρήσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις όπου μιλάμε για καθαρά εκτελεστικές ε, δραστηριότητες ε, μπορεί να συζητηθεί αυτή η πτυχή της αυτονομίας και να αναθεωρηθεί ενδεχομένως. Η εκθέση του συναδέλφου Σόπλινγκ περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέρουσε προτάσει. Δεν προλαβαίνουμε τώρα, αλλά αξίζει τον κόπο να τη συζητήσουμε σε βάθος. Σίγουρα μια καλή πρόταση είναι αυτή η ετήσια συζήτηση που θα οργανώνεται μέσω της δικής μας Επιτροπής και που στη συνέχεια θα συνεχίσετε στο Κοινοβούλιο εξετάζοντας τα συνολικά ζητήματα της λειτουργίας ε, και της ποιότητας ε, της εκτέλεσης από αυτούς τους οργανισμούς ε, της δουλειά τους δηλαδή αναμφίβολα η πιο σημαντική πτυχή του ελέγχου αυτή τη στιγμή εκ μέρους του Κοινοβουλίου είναι η, απαλλαγή, η δημοσιονομική απαλλαγή και η έγκριση των προληπτικών προπολογισμών. Ο έλεγχός μας ωστόσο επικεντρώνεται υπερβολικά σε αυτές μόνο τις πτυχές, οι οποίες να μένουν σημαντικές, αλλά όσον αφορά την εφαρμογή αυτή καθεαυτή των ευρωπαϊκών ε, νόμων, από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Πολύ συχνά οι πληροφορίες που μας έρχονται είναι πιο κατακριματισμένες. Πολύ περισσότερο μάλιστα. Και ανεπαρκείς. Κάποια γενική λοιπόν συμφωνία η οποία ενδεχομένω θα καθορίζει και θα ταξινομεί τους οργανισμούς ε, αναομάδες διαφόρων χαρακτηριστικών όπου θα ορίζεται και τι είδου εκθέσεις ε, δραστηριοτήτων θα πρέπει να καταθέτουν οι οργανισμοί στο Κοινοβούλιο και στα ελεγκτικά όργανα γενικότερα. Πιστεύω και αυτό παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον. Όπως είπα λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση. Περιλαμβάνει πολλές προτάσεις, πολύ καλές, ε, αποτελούν καλή βάση. Ελπίζουμε πριν το τέλος της θητείας να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε πιο καλά τις προτάσεις ξεχωρίζοντας τις προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση και τις προτάσεις ε, που απαιτούν τροποποίηση του συνθήκης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μερσέδες. Τους φιλελευθέρους γιατί αποσιάζουν οι συντηρητικοί είτε Παγάσα Ορτοντούα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς Πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετικό το έργο που κάνετε κύριε Σιγητά σε όλο αυτό το θέμα. Και εγώ έχω επισκεφθεί αποκεντρωμένους οργανισμούς και είδα και τις διαφορές που έχουν μεταξύ τους. Έχουν πολύ μεγάλη εξειδικευσή και ανάγκη ανεξαρτησίας για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στις προκλήσεις ε, και στο έργο για το οποίο έχουν δημιουργηθεί το θέμα της ε, λογοδοσίας και της ε, διακυβέρνησης ε, μπορεί να είναι γενικά, αλλά δεν μπορούμε να τους βάλουμε και ένα στενό κορσέ για να μην μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, δουλειά για την οποία συστήθηκαν. Συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι σε περίπτωση αναθεώρησης των συνθηκών θα πρέπει να ορίζονται καλύτερα οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί γενικότερα. Αλλά επιμένουμε στο γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη, ε, πρακτική ανάγκη να μπορούν να δουλεύουν. Να μην είναι ε, στήρα αυτή η προσπάθεια υπερβολικά γραφειοκρατική και στραγγαλιστική για να μην μπορούν να κάνουν την ειδική δουλειά για την οποία δημιουργήθηκαν. Και επίσης ε, τα άλλα που λέτε για τη διακυβέρνηση, για τη λογοδοσία, για τη διαφάνεια είναι πολύ σωστά. Βεβαίω, αν αυξηθούν οι μηχανισμοί που υπάρχουν, και υπάρχουν και κάποια που επιβάλλουμε εμείς στον εαυτό μας, αλλά θα πρέπει να προετοιμαστεί και το προσωπικό ε, και να προσαρμοστεί ε, ε, ο προϋπολογισμός των οργανισμών. Αλλιώς θα τους κατακλείσουμε, θα τους πνίξουμε με διάφορες διοικητικές υποχρεώσεις και δεν θα μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Και δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Γενικά έχω να προσθέσω το εξής. στις επιτροπές ΛΥΜΠΕ, ΠΑΝΑ και ΤΕΡ είδα κάποιους οργανισμούς που ήταν ε, πάντα πρόθυμοι να συνεργαστούν με το κοινοβούλιο και όταν τους ζητούσαμε να έρθουν να λογοδοτήσουν ήρθαν να λογοδοτήσουν και επιζητούν και επιθυμούν ε, περισσότερη επαφή μαζί μας και μεγαλύτερη σύνδεση για να μην ε, αποξενωθούν από την κοινοβουλευτική δουλειά και τις σχέσεις με τους βουλευτές. Πολλές φορές λοιπόν όταν αναλύουμε τους οργανισμούς αυτούς δεν συνειδητοποιούμε ότι καμιά φορά υπάρχουν μερικά ζητήματα τα οποία οφείλονται σε εμά. Δεν αξιοποιούμε πλήρως ως κοινοβούλιο ή ως μονομένοι βουλευτές όσα έχουν να μας προσφέρουν οι οργανισμοί αυτοί να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Φυσικά θα συνεργαστούμε με τον εισηγητή που είναι πάρα πολύ σοβαρός και επιμελής στην έκθεσή του και θα κάνουμε και τροπολογίες που θα σας ε, αναλύουν τη θέση των φιλελευθερών. Ευχαριστώ πολύ. Από τους Πρασίνους, ο κύριος Μαξ Άντερσον. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή την εισηγήτρια. Τον εισηγητή. Η πράσινη είναι πολύ θετικά προσκύμενη στην έκθεση αυτή. Όλα μας φαίνονται εντάξει και μας αρέσει ιδιαίτερα η πρόταση για, την, ε, για τις διοργανικές συμφωνίες κάθε πέντε χρόνια. Αλλά να κοιτάξουμε λίγο περισσότερο την διατύπωση σχετικά με τη διαφάνεια, διότι υπάρχει μία κάποια ασάφεια και βέβαια μας αρέσει η κατεύθυνση της εκθέσης, όμως ε, νομίζω πως χρειάζεται να πάμε λίγο πιο πέρα και να είμαστε περισσότερο σαφείς ε, σχετικά με το πόση διαφάνεια θέλουμε σε αυτές τις υπηρεσίες. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα χαρώ πολύ να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Οι άλλες πολιτικές ομάδες απουσιάζουν. Να πω προσωπικά το εξής μόνο σύμφωνα με την εμπειρία μας. Υπάρχει τρόπος να συνεργάζεται μια κοινοβουλευτική επιτροπή στενά με έναν οργανισμό και ταυτόχρονα να τον ελέγχει. Και αυτός ο τρόπος ποιος είναι, να εξασφαλίσουμε ο διευθυντής του οργανισμού να διορίζεται με τη συμφωνία του Κοινοβουλίου θα μπορούσαμε να το δρομολογήσουμε αυτό χωρίς αναθεώρηση των συνθήκων ή χωρίς αναθεώρηση του καταστατικού των οργανισμών αυτών. Έχουν επικρατήσει κάποιες συνήθειες, ας πούμε, στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Όλοι οι οργανισμοί που εξαρτώνται, κυρίως οι τρεις ρυθμιστικές αρχές, η Τραπεζική Αρχή, η Αρχή των Ασφαλίσεων και των Χρηματαγορών, έρχονται στην Επιτροπή ΕΚΟΝ κάνει ακροάσεις ε, βέβαια άτυπες με τους υποψηφίους και γίνονται και συστάσεις άτυπες στο Συμβούλιο. Και από εκεί και πέρα το Συμβούλιο επιλέγει και νομικά μπορεί και να διορίσει ε, αλλά γίνεται και άλλη ακρόαση επίσημη αυτή τη φορά του υποψηφίου που ε, ήταν ο επικρατέστερος στην οικονομική και νομισματική. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν ο διευθυντής του οργανισμού έρχεται για να λογοδοτεί τακτικά ε, στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Υπάρχει μια τέτοια σχέση που έχει σφυριλατηθεί και μου φαίνεται αρκετά γόνιμη. Έτσι μπορεί και το Κοινοβούλιο να έχει μια εικόνα για τον προσανατολισμό και την κατεύθυνση που παίρνει ο οργανισμός και να είναι και προς την κατεύθυνση του Κοινοβουλίου φυσικά. Ε, δεύτερον, παρακολουθώ και την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ε, την προηγούμενη θητεία μου και πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Γιατί διαπίστωσα εκεί. Δεν είχαμε ποτέ βρει την καλή λύση για να δουλέψουμε ε, στα σχέδια προϋπολογισμών των ε, οργανισμών. Παρίστατη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπό της. Όπως άριστα εξήγησε ο εισηγητής, υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισμοί αποκεντρωμένοι που είναι πάρα πολύ διαφορετικοί και ε, από την εμβέλεια των εξουσιών τους, από το προσωπικό που έχουν, από τους πόρους που έχουν για τους οικονομικούς, από την αρχαιότητά τους ακόμα, γιατί υπάρχουν οργανισμοί που συστήθηκαν πρόσφατα και είναι σε φάση σταδιακής αύξησης των δραστηριοτήτων και του προσωπικού για να πάρουν μια κανονική ταχύτητα και υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί που είναι πιο παλιοί και έχουν μπει σε μια ρέγουλα. Και κάθε φορά που εξετάζουμε το σχέδιο προϋπολογισμού για το επόμενο οικονομικό έτος, εκείνοι που ασχολούνται με τον προϋπολογισμό τείνουν να τις βάλουν όλες στο ίδιο τσουβάλι. Ας πούμε, 1% οριζόντια μείωση των λειτουργικών δαπανών ή οροφή όλων των λειτουργικών δαπανών για όλους τους οργανισμούς. Αυτό δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό. Σίγουρα χρειάζεται και προποθέτει αυτό καλύτερο συντονισμό μεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισμών και των άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών του Κοινοβουλίου που παρακολουθούν τις εργασίες των ε, αποκεντρωμένων οργανισμών. Αλλά αυτό είναι θέμα εσωτερικής οργάνωσης του Κοινοβουλίου, αλλά μπορεί και πέρα από αυτό να μας απασχολήσει και να προβληματιστούμε και να συζητήσουμε και με τα άλλα θεσμικά όργανα. Παρίσταται λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Χένινγκ Κλάους. Θεμηματάρχης των ε, διοργανικών σχέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Thank you. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έκθεση αυτή, είναι εξαιρετική και ο κύριος Σόφλιν εργάστηκε πολύ καλά. Επίσης, ε, θεωρούμε πως και η δουλειά του κύριου Φως είναι πάρα πολύ καλή. Υπάρχουν κανόνες διακυβέρνησης και όλοι αυτοί έχουν αποτελέσματα. Να σας υπενθυμίσω σύντομα ότι η κοινή προσέγγιση του 2012 ήδη αποτελεί διοργανικό κείμενο. Δεν είναι ακόμα διοργανική συμφωνία όπως προβλέπει η συνθήκη, όμως είναι ένα κείμενο το οποίο ε, έχουν διαπραγματευτεί τα τρία θεσμικά όργανα και μάλιστα με δύσκολες διαπραγματεύσεις. Το αποτέλεσμα είναι λοιπόν αυτή η κοινή προσέγγιση και είναι ό,τι ήταν εφικτό εκείνη την εποχή. Γι' αυτό είναι ένα πάρα πολύ ευέλικτο κείμενο, διότι συμπεριλαμβάνει όλη την, ε, όλο το εύρος των οργανισμών και εξετάζει όλες ε, τις ε, περιπτώσεις που είχαν προκύψει. Γι' αυτό και παρέχει πολύ ευελιξία και είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται τακτικά από τον νομοθέτη. Τώρα, έξι χρόνια αργότερα έχουμε μία έκθεση η οποία δεδομένη της ε, λοιπού συμμόρφωσης ε, των ε, οργανισμών με την κοινή προσέγγιση και δεδομένων των εμπειριών που έχουμε αποκτήσει σχετικά με την εποπτεία Προτείνει λοιπόν η έκθεση μία πλήρη αξιολόγηση. Να σας υπενθυμίσω βέβαια ότι η έκθεσή σας ασχολείται μόνο με θέματα δημοκρατικού ελέγχου, καθώς και η μελέτη του καθηγητή κ. Βος. Υπάρχουν και άλλα θέματα όμως, τα οποία δεν εξετάζει αυτή η Επιτροπή και το αναφέρω αυτό διότι παρόλες τις ελλείψεις σχετικά με τη συμμόρφωση υπάρχει ήδη μεγάλη προστιθέμενη αξία. Για παράδειγμα, η εναρμόνιση ε, της νομοθεσίας σχετικά με τις αρμοδιότητες των ε, διευθυντών, οι συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και ε, υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δεν είμαστε και απόλυτα πεπισμένοι με αυτήν την στενή σχέση ανάμεσα στη, στα κράτη-μέλη και τις έδρες των οργανισμών αυτών. Θα θέλαμε να ανταποκρίνονται περισσότερο τα κράτη-μέλη στις ανάγκες των οργανισμών αυτών σε ό,τι αφορά τις διεθνείς τους δραστηριότητες. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτήν την πλήρη αξιολόγηση, το επόμενο στάδιο δηλαδή, που είναι και πιο φιλόδοξο, έχουν γίνει, ε, ε, υπάρχουν μάλλον ε, τέτοιες προβλέψεις στις ιδρυτικές πράξεις των οργανισμών αυτών. Δέκα αυτή τη στιγμή βρίσκονται εν εξελίξη και παρά ορισμένα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι θα θέλαμε ακόμα περισσότερα στοιχεία. Θα προτιμούσαμε πρώτα να ολοκληρωθούν αυτά τα δέκα νομοθετήματα σχετικά με τις ιδρυτικές πράξεις και μετά να κρίνουμε από αυτά πώς θα προχωρήσουμε. Το είπα στην αρχή. Η διοργανική συμφωνία βάσει συνθήκων δεν σημαίνει αυτόματα και καλύτερη συμμόρφωση. Καταρχάς υπάρχει ε, η νομοθεσία και καλύτερη νομοθεσία, έτσι ώστε όλοι οι οργανισμοί της Ένωσης ε, να διακρίνονται από αυτήν την συμμόρφωση. Αλλά να πω και κάτι σχετικά με τον προϋπολογισμό, κύριε Λαμασούρ στο προηγούμενο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο υπήρχε υποχρέωση σε ό, για όλα τα κρατη να υπάρξουν περικοπές ε, οριζόντιες ε, της τάξης του 5% για όλους τους οργανισμούς. Υπάρχουν όμως και ορισμένες ε, περιπτώσεις ε, οργανισμών που ανέλαβαν πρόσθετα καθήκοντα που χρειάζεται ε, κάποιο χρόνο γιατί ήταν ε, οργανισμοί και υπηρεσίε που είχαν δημιουργηθεί πρόσφατα. Αυτός ο γενικευμένος οριζόντος χαρακτήρας δεν υπάρχει πια. Ελπίζω να μην ε, χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ξανά στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και μπορούμε φυσικά να κάνουμε εξαιρέξεις, αλλά αυτό ε, περιέχει πολλές από το που θα συζητήσουμε στη συνέχεια στην περίπτωση αυτή μπορούμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ομαδοποίησης ορισμένων οργανισμών για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνται. Θα μπορούσαμε να τις ομαδοποιήσουμε ανατομία πολιτικής, για παράδειγμα. Ε, και δεν αναφέρομαι εδώ σε θέματα λογοδοσίας, υποβολής εκθέσεων, σύστασης, ε, σύνθεσης μάλλον διοικητικού συμβουλίου κτλ. Αυτά σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Τώρα, φυσικά, ε, μπορώ να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανταποκριθεί στο αίτημα του Κοινοβουλίου που εγκρίνατε στην ολομέλειά σας και για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος εισηγητής, αν θέλει, για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα πω ιδιαίτερα συμπεράσματα, αλλά θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν ε, στη συζήτηση. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και στις τροπολογίες. Ε, με ερώτηση που ήθελα να κάνω, ε, είπα σαφώς στην εισαγωγή μου ότι δεν είμαι Βίνος, δεν είμαι υπέρ της, του κεντρικού ελέγχου. Θέλω να βρούμε μια καλή ισορροπία με επαρκή εποπτεία, αλλά διατηρώντας ε, την αυτονομία των οργανισμών. Και δεν είπα ποτέ ότι είναι εύκολο. Θέλω να ευχαριστήσω με ευγνωμοσύνη την ε, ε, Κομισιόν για τις πληροφορίες, πολύ ενδιαφέρουσες. Μ' αρέσει η ιδέα ενός διοργανικού κειμένου. Δεν μιλάμε για διοργανική συμφωνία, για κοινή προσέγγιση είναι καλό να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία διοργανική, πολύ χρήσιμη θα ήταν πιστεύω. Θέλω να ευχαριστήσω τον εκπροσωπό της Κομισιόν για όσα προσέθεσε. Ήταν πολύ πολύτιμες πληροφορίες αυτές για την έκθεση αυτή. Και ελπίζω πραγματικά ότι η Ολομέλεια θα το υιοθετήσει κάπου στις αρχές του νέου έτους. Οπότε θα υπάρχει το κείμενο έτοιμο για να το δουλέψει το νέο κοινοβούλιο. Αυτό προσπαθώ να επιτύχω με αυτή την έκθεση. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ρίτσαρντ, συγγνώμη, ένα πράγμα δεν κατάλαβα από αυτά που συνοψίσατε. Μιλήσατε για διοργανικό κείμενο που δεν είναι συμφωνία. Τι είναι τότε, ε, διοργανική διαφωνία. It's a nice idea. Καλή ιδέα, αλλά απλά αναφέρομαι σε αυτά που είπε η Επιτροπή δεν υπάρχει διοργανική συμφωνία, αλλά διαπραγματευτήκαμε ένα κείμενο το οποίο αποτέλεσε την κοινή μας προσέγγιση. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε άτυπο. Δεν είναι διαφωνία απαραίτητα, απλά δεν έχει κάποια ισχυρή νομική διοικητική βάση. Η εντύπωση που έχω είναι ότι υπάρχει η κοινή προσέγγιση, αλλά φυσικά υπάρχουν διαστάσεις απόψεων. Σίγουρα δεν υπάρχουν σοβαρές παρεκκλήσεις, αλλά εκεί τίθεται και ε, το ζήτημα της διακυβέρνησης φυσικά. Κάποιο μνημόνιο δηλαδή συνεννόηση, κάτι τέτοιο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ όλους όσοι ε, συμμετείχαν στη συζήτηση και ειδικότερα τον εισηγητή. 17 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών, εξέταση των τροπολογιών στην Επιτροπή 22 Ιανουαρίου. Προβλέπεται η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΑΦΚΟ 29 Ιανουαρίου και έγκριση στην Ολομέλεια είτε το Φεβρουάριο είτε στην πρώτη σύνοδο του Μαρτίου. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πολύ ωραία. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε εξαντλήσει την πρωινή ημερήσια διάταξη εκτό από τι ψηφοφορίε, οι οποίε ψηφοφορίες όμω έχουν προβλεφθεί να λάβουν χώρα σε μισή ώρα από τώρα. Οπότε σα προτείνω να διακόψουμε μέχρι τις 45. 12 παρατέταρτο. Παρακαλώ να είστε εδώ ακριβώ και παρακαλώ οι βοηθοί των ομάδων να βεβαιωθούν ότι θα έχουμε απαρτία επαρκή για να ψηφίσουμε τα σημαντικά αυτά κείμενα σε μισή ώρα από τώρα στις 12 παρατέταρτο. Η συνεδρίαση αναστέλλεται.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE Είναι Mes chers collègues. Αγαπητοί συνάδελφοι. Ναι. Il est 11h45, nous commençons la... Είναι 12 παρατέταρτο και είχαμε πει ότι θα αρχίσουμε τις πληροφορίες. Από ό,τι φαίνεται έχουμε και απαρτία. Vous avez tous votre liste de vote. Je propose... Έχετε όλοι τον κατάλογο ψηφοφορίας σας. Να κάνουμε μια δοκιμή για να δούμε αν λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα. Αρχίζει τώρα. βότε, βότε. voté. Ψηφίσατε. Voilà. για 17 βοτών. 17 ψήφισαν. Για 17 βοτών και il n'y a pas 17 ψήφισαν. Και δεν υπάρχει υπεράριθμος από το ΕΛΚ για αλλαγή. Δεν υπάρχει, υπάρχει, μην βγάζετε. No, no. No, no. It's the case when Elmar Brock is uh, uh, present, but it's... Όταν είναι εδώ ο Μπροκ πάντα περισσεύει ένας από το ΕΛΚ, αλλά τώρα είμαστε εντάξει. <laughs> okay. Bien. Alors, tout le monde a sa liste de vote, tout le monde est prêt. Λοιπόν, πάνε έτοιμοι, πάμε. Έκθεση Ρίτσαρτ Κόρμπετ. Θέλει ο να πει τίποτα. Όχι. Προτιμάει να σιωπήσει. Block vote παριθμόν 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν κρίνεται. Η τροπολογία 5 του Ρίτσαρτ Κόρμπετ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν κρίνεται. Η τροπολογία 9 του ιδίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 του ιδίου με προφορική τροπολογία αρκετά μακροσκελή που δεν χρειάζεται να τη διαβάσουμε γιατί τη βλέπετε εδώ γραμμένη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 71 των πρασίνων Καταπίπτει. Διότι εγκρίναμε την 5. Προχωρούμε. 72. Επίσης κατέπεσε. 73. Το αυτόν. Διότι εγκρίθηκε η τροπολογία υπαριθμών 10. Ε, block vote υπαριθμών 2. Βε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, ομαδοποιημένη πάλι παριθμό 3. Βε. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά στο τσεκάρουμε για καλό και για κακό. Α, τώρα περσέβει ένα του ΕΛΚ. Μάλιστα, τον βρήκαμε τον υπεράριθμο. Καλά, δεν θα ψηφίζω εγώ λοιπόν. Ε... No, no, no, I, I my Να έβγαλα εγώ την κάρτα μου, μην βγάλετε τώρα όλοι του ΕΛΚ. Ως πρόεδρος δεν θα ψηφίζω. Λοιπόν, 21 είμαστε από το ΕΛΚ. Καλώς. 21 ε, ε, σύνολο. 13 ε, υπέρ, 8 κατά εγκρίνεται. Και προχωρούμε. Στην τροπολογία υπαριθμών 74, το πρώτο μόνο τμήμα όμως, γιατί τα δύο επόμενα έχουν καλυφθεί. Το δεύτερο καταπίπτει και το τρία... Με το 3 τι γίνεται. Καλά, ας δούμε πρώτα το πρώτο. Ψήφι υπέρ. Κατά. Τα μαμούθ είναι αντίθετα, οπότε απορρίπτεται. Και το, το δεύτερο τμήμα έχει καταπέσει, το τρίτο τώρα έχει νόημα. Έχει λένε. Ο εισηγητής τι λέει. Έχει νόημα να ψηφίσουμε το τρίτο τμήμα χωρίς τα δύο πρώτα. Ο κύριος Κόρπετ Έτσι και πιστεύω ότι θα απορριφθεί. Οπότε ας την ψηφίσουμε. Εντάξει. Η ένδειξη μαζοχισμού ζητάει ο εισηγητής να ψηφίσουμε μια τροπολογία ελπίζοντας να καταψηφιστεί. Μα μιλώ για την 74, δεν είναι δική μου η τροπολογία, λέει ο κ. Κόρμπετ. Υπέ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ερχόμαστε τώρα στην τροπολογία του εισηγητού που είναι 16, είπε. Και contre. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17, είπε. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 20 έχει αποσυρθεί. 4, ομαδική ψηφοφορία, είπε. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 19 εκτός από την παράγραφο 2 υπέρ. Αποχές εγκρίνεται. 65 δεν είναι παραδεκτή. 19, τώρα την παράγραφο 2 στη 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66 και 67 καταπίπτουν. Αφού εγκρίθηκε 19-2. Ερχόμαστε στη συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Α, αυτό θέλει έλεγχο. Και εγώ δεν θα ψηφίσω. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. 11 υπέρ, 10 κατά. Αυτά είναι. Μήπως έπρεπε να ψηφίσω. Να είχα ψηφίσει. Τι να κάνουμε. Αν ήμασταν στη Γαλλία κάτι θα γινότανε. Ε, συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69 καταπίπτει και 70, 75 έχει αποσυρθεί. Η επόμενη ψηφοφορία των 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 του Κόρμπετ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 με προφορική τροπολογία που λέει ότι θα οργανώνεται στη δεκτήρια του Κοινοβουλίου υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το ΕΛΚ είναι μόνο αντίθετο σε αυτή την τροπολογία. Ε, τροπο, ε, ψηφοφορία 6, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26. Το εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Block vote παριθμών 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και ερχόμαστε στην τροπολογία 34 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35. Τώρα εδώ έχουμε μια σειρά τροπολογιών από την 35 έως την 43 που είναι όλες του Ρίτσαρτ Κόρμπετ. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Θαυμάσια, τέλεια. Λοιπόν, 35 με 43, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Και φτάσαμε στην τροπολογία Επειδή κάποιες καταπίπτουν, 77, 78, 82, 79, 80 καταπίπτουν και 81 84-85 επίση. 83 καταπίπτει και αυτή. Η 86 ναι και 87 και η 88 δεν είναι παραδεκτή. Βότ, μπλοκ, 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα Πάμε στην επόμενη αιμαδική ψηφοφορία, την 9, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 51 τώρα, υπέρ κατά δις αποχές εγκρίνεται ομόφωνα. Η τροπολογία 93, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 94, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 καταπίπτει. Η 95 μπορεί να ψηφιστεί ε, ως προσθήκη στην 53 υπέρ της 95. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η Άλτε έχει απομονωθεί σφόδρα. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η ομαδική ψηφοφορία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 98 υπέρ μερικοί είναι υπέρ κατά η πλειοψηφία αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά και οι σοσιαλιστές τίποτα αποχή θα ψηφίσετε αποχή ε, να ψηφίσουμε γιατί απέχουν οι σοσιαλιστές. Όχι, ε, ε, ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίστε, ψηφίστε, ψηφίστε. Δεν σας βλέπω Χαλαρίστε. είστε, ξυπνήστε. 21. 5 υπέρ, 10 κατά και 6 εποχές. Απορρίπτεται αυτό. Και ποια ήτανε? Η 99. Απερίφθη. 100. Έχει ψηφοφορία κατά τμήματα που ζήτησαν οι φιλελεύθεροι να ψηφιστούν χωριστά οι λέξεις να μεταφράζονται σε, στις ε, επίσημες γλώσσες και, και τι και στις ανεπίσημες, υπέρ, κατά, αποχές. Οι μεγάλες ομάδες κερδίζουν και απορρίπτεται. Επίσης, ομαδική ψηφοφορία 11 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 101 καταπίπτει, 102 και 103 μαζί έχει και προφορική τροπολογία που ζητάει ο συγητής για να διαγραφεί η λέξη ολομέλεια. Υπέρ κατά της διαγραφής αυτής εποχές εγκρίνεται. Με 104. Προφορική τροπολογία. Ορίστε, Ρίτσαρτ. Νομίζω ότι ψηφίσαμε να βγει η λέξη πλήναρη αλλά πρέπει να ψηφίσουμε και τις υπόλοιπες τροπολογίες, όχι μόνο την προφορική. Πολύ εύστοχο το σχόλιο σας κύριε Σιγητά μου. Εγώ πταίω. Άρα ψηφίζουμε τις δύο τροπολογίες ε, χωρίς την λέξη ολομέλεια. Υπέρ. Το ΕΛΚ. Σε ποια τροπολογία είμαστε, Πρόεδρε. 103 και 102 είναι οι ίδιες. Χωρίς τη λέξη ολομέλεια. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 104. Έχουμε προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Τα μεγάλα τάγματα το πέριψα. 105 ψηφίζεται έτσι γιατί δεν εγκρίθηκε το 104 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται 106 υπέρ όχι Πού πάμε τώρα Στην 61 Υπέρ Κατά Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Με προφορική τροπολογία στην παράγραφο 2 για το σχέδιο απόφασης. Μα μου λένε ότι αν απορριφθεί... Ε, όχι, τίποτα, τίποτα. Εντάξει, προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα τώρα δεν χρειάζεται να ξαναψηφίσουμε τη γραπτή ε, ε, τροπολογία δεν υπήρχε, ήταν μόνο η προφορική. Τελική ψηφοφορία τώρα, ονομαστικά και ηλεκτρονικά προφανώς. Εγώ δεν ψηφίζω, λέει ο Πρόεδρος. Πέρας. Ομόφωνα. 21 υπέρ. 0, ε, κατά 0 αποχές. Et donc, euh, Καθώς λοιπόν το Κροατήριο είναι πιο πολυπληθές από ό,τι σήμερα το πρωί, να επαναλάβω την πρόταση να ψηφίσουμε ένα ψήφισμα ώστε ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ να γίνει Ευρωπαίος πολίτης διαβίου στην ε, δυστυχή περίπτωση όπου το Brexit ε, υλοποιηθεί. Ρίτσαρτ, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρο, για το πολύ ευγενικό σα σχόλιο. Πρώτα απ' όλα, ήθελα να ευχαριστήσω όλου του ε, συναδέλφου και φυσικά και τα μέλη τη ομάδα εργασία που έγιναν και σκιώδη μου, γιατί η δουλειά αυτή δεν είναι μόνο δική μου. Ήταν συνεργατική δουλειά μεταξύ όλων των ομάδων που βρήκαν μια επικοδομητική συνένεση για να βελτιώσουμε τους κανόνες μας, να εργαζόμαστε πιο αποτελεσματικά, πιο αποδοτικά, πιο, με μεγαλύτερη διαφάνεια και ελπίζω αυτή η ομοφωνία επί όλων των σημείων να επαναληφθεί όταν θα ψηφίσουμε στο, σε ολόκληρο το κοινοβούλιο, ολόκληρο το κοινοβούλιο, όποτε γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Είμαι βέβαιος ότι όλοι οι συντονιστές των ομάδων θα μεριμνήσουν ώστε να επαναληφθεί η ίδια ομοφωνία και μεταξύ των 751 συναδέλφων μας. Περνάμε τώρα στην έκθεση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των ε, ευρωεκλογών. Ε, θέμα το οποίο μας αφορά ιδιαίτερα. Έχουμε πρώτα απ' όλα μια τροπολογία ΛΥΜΠΕ 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. απορρίπτεται. Τροπολογία 1 του κυρίου Ντουραν, ε, υπέρ. Πράσινη, κατά. Όλοι οι υπόλοιποι, όχι μόνο η πράσινη και η γκουε. Ποιο είναι κατά ε, πλειοψηφία. Απορρίπτεται 2 ταυτόσημες, 2 και λίμπε 2, υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνονται. 3 Γανζέλ, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 4 αντιράν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 Βίλαντ και Μπρέσο η μεγάλη συμμαχία υπέρ κατά ο μεγάλος συνασπισμός ε, εγκρίνεται Λίμπε 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 Σελίμοβιτς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 Αντιράν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 Αντιράν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 Αντιράν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Λίμπε 4 και 10 Σελίμοβιτς είναι ταυτόσιμες όχι Τότε λίμπε 4. Η εισηγητής τι θέλει. Είναι κατά ο εισηγητής. Γιατί δεν είναι στο κατάλογο ψηφο Δεν είναι. Λοιπόν, η 10. Η λίμπε 4, συγγνώμη, ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10, Σελίμοβιτς υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11, Ντιραν, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 12 Βίλαντ και Μπρέσο υπέρ κατά αποχ... α... αποχές εγκρίνεται Λίμπε 5 και 13 του Σελίμοβιτς είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Λίμπε 6 και 14 Σελίμοβιτς ταυτόσιμες επίσης υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 τη, μεγάλου συνασπισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται εγκρίνεται τελική ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία ονομαστική Να βλέπω ψηφίζουμε καλύτερα μα τέλος ψηφοφορίας 21 υπέρ, 0 κατά, 0 αποχές. Alors, il faut maintenant voter sur la... Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε για την πρόταση έναρξης οργανικών διαπραγματεύσεων. Διανατασχερός είναι η ίδια πλειοψηφία υπέρ, κατά αποχές η ίδια ομοφωνία είναι. Ah, mais euh, Madame le rapporteur, Merci. le co-rapporteur, ε, ήθελα ε, και εκ μέρους του να ευχαριστήσω άπαντες. Πολλές από τις τροπολογίες μας ήταν διότι αποφασίσαμε να, να διατηρήσουμε την πρόταση αυστηρά στις, ε, όσον αφορά τις ευρωεκλογέ, να μην το επεκτείνουμε στα κόμματα. Υπάρχουν, θα έχουν και άλλες ευκαιρίες, αλλά για να έχουμε μια συμφωνία γρήγορα και να τεθεί σε ισχύ πριν από τις ευρωεκλογέ, έπρεπε να περιοριστούμε σε αυτό. Γι' αυτό το λόγο, μεταξύ άλλων, πολλές προτάσεις δεν έγιναν δεκτές. Ευχαριστώ. Bien. Alors, Euh, Ωραία, για την τελευταία ψηφοφορία. η πρόεδρος Ντανούτα Χούμπνερ που είναι και η συγγήτρια ε, για αυτή την έκθεση τροποποίησης του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ώστε να ληφθεί υπόψη αυτό το δυστυχές ε, σενάριο του Brexit που είναι μια δυνατότητα με πιθανότητα ζητά απλοποιημένη διαδικασία χωρίς τροπολογίες σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 αν συμφωνείτε λοιπόν χωρίς ψηφοφορία θα εγκρίνουμε τα συμπεράσματα της έκθεσης της κυρίας Φιμπνερ χωρίς ψηφοφορία, χωρίς τροπολογίες. Pas δεν αντιτίθεται κανένας, όλοι συμφωνούν. Σήμερα το πρωί όλοι συμφωνούν. Να είναι καλά ο Νικόλας, ο Άγιος Νικόλαος. Διακόπτε λοιπόν η συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε στις 2 ακριβώς. Καλή σας όρεξη.